So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte auf die Plätze. Καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι. Θα μπορούσαμε ίσως να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό, γιατί έχει πολύ γρασία μέσα στην αίθουσα. Λοιπόν, δεν έχουμε αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Προχωρούμε στις ανακοινώσεις. Έχουμε όλες τις γλώσσες στη διάθεσή μας. Έχουμε και ε, τα... Ε, ταξίδια στην Ιρλανδία Κοπενχάγη 28-29 Απριλίου έγινε... Όχι, αυτά είναι ταξίδια που έγιναν. Έχαμε και μια ομάδα 26 επισκεπτών σήμερα μετά από πρόσκληση της κυρίας Γκροστέτ. Θα έρθουν στις 2.30 και θα μείνουν μέχρι τις 3.30. Ε, μετά για τους τριμερείς διαλόγους, ε, για τα ε, αέρια... Έφε, Έχουμε μια κρόαση από το απόγευμα. Το EBS. Για το EBS αύριο θα γίνει ε, τριμερής διάλογος για τα καπνά επίσης. Ο δεύτερος έγινε στις 12 Νοεμβρίου και ο επόμενος τριμερής διάλογος θα γίνει στις 9. Από τις 9, όχι, 9 με 12 Δεκεμβρίου λέει εδώ. Τι τριμερής διάλογος τριμερος θα είναι αυτός με το Συμβούλιο και τις κλινικές δοκιμές στις 4 Δεκεμβρίου και τον τελευταίο στις 12 Δεκεμβρίου. Χθες είχαμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο για το διοξίδιο του άνθρακα και τα αυτοκίνητα έκθεση Ούλμερ και μπορούμε να πούμε ότι η συμβιβαστική λύση είναι αποδεκτή από το Κοινοβούλιο 5% των οχημάτων θα μπορούν επί 365 μέρες να έχουν μεγαλύτερη τιμή από την προβλεπόμενη 94 γραμμάρια. Όλα τα άλλα παραμένουν όπως είχαν κατά τον τριμερή διάλογο του Ιουνίου. Οπότε δώσαμε τη μάχη μας εκεί και πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τον εισηγητή που ως ομάδα έκαναν πολύ καλή δουλειά. Ο Μάριο Πυρίλο ε, ήταν ο Σκιώδης και ε, σας ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε με τα πρακτικά από 10 Οκτωβρίου, 17 και 24 Οκτωβρίου υπάρχουν τα πρακτικά, δεν υπά... αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις γίνονται δεκτά και αρχίζουμε με την έκθεση του Σκιώδους που τον αναφέραμε πριν από λίγο αλλά τώρα είναι κανονικός εισηγητής, μιλώ για το σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη και την έκθεση Πυρίλο και ο Μάριο Πυρίλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε νομίζω όλοι όσον αφορά τους απαραίτητους επίσημους ελέγχους για την ασφάλεια των προϊόντων μας και για τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας. Ε, αυτοί οι έλεγχοι βοηθούν στο να διατηρείται υψηλή η ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων στο διεθνές επίπεδο και βοηθούν την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξάγει προς τρίτες ε, χώρες και βάσει των αυστηρών ε, προτύπων ασφαλείας που προσθέτουν προστιθέμενη αξία σε σχέση με άλλες γεωγραφικές περιοχές. Ο κανονισμός τον οποίο είμαι εισηγητής αποτελεί κομμάτι του νομοθετικού πακέτου που δημοσίευσε το Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντάσσεται στην ε, στρατηγική από το σπόρο μέχρι το τραπέζι έτσι ονομάζεται η οποία καλύπτει όλους τους κανόνες για την ε, δημόσια υγεία ώστε να διασφαλίζεται ότι τα τρόφιμα παράγονται και εξάγονται δεν είναι επιβλαβή πρόταση κανονισμού επεκτείνεται επίσης και στους επίσημους ελέγχους ε, για τα φυτά που εξαιρούνταν προηγουμένως στο κανονισμό 882 του 2004. Υποστηρίζω την πρόταση της Κομισιόν διαταπλοποιεί τη χρήση πιο συνεκτικών ελέγχων, αναλογικών με τους κινδύνους και δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο αναρμονισμένο για τις διαδικασίες ελέγχων. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε ώστε να ορίσουμε σαφείς κανόνες για να περιορίσουμε τα προβλήματα που είχαμε μέχρι σήμερα και τα οποία οφείλονταν κυρίως στις ε, εθνικές ερμηνείς που συχνά αποτέλεσαν την αιτία ανομοιόμορφης εφαρμογής του κανονισμού που ισχύει. Πριν μπω στις λεπτομέρειες της δικής μου έκθεσης, επιτρέψτε μου να κάνω μια εισαγωγή, υπενθυμίζοντας ότι πριν, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πραγματική ανταλλαγή απόψεων. Γι' αυτό τον λόγο το έγγραφο αυτό θεωρείται περισσότερο σχέδιο παρά τελικό έγγραφο και σίγουρα δεν είναι ολοκληρωμένο. Σίγουρα μπορούμε να παρέμβουμε και να συμπληρώσουμε το κείμενο και δεδομένων επίσης και των παρατηρήσεων που θα ακούσουμε στη σημερινή συζήτηση. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε ορίσει συγκεκριμένε συχνότητε ε, για τους ελέγχους και έτσι βρισκόμαστε πάντα ενώπιον ε, διαφορών μεταξύ κρατών μελών. Στον τομέα της τυροκομείας ε, έχουμε χώρες όπου ανούν χώρα κάθε 10 χρόνια ενώ σε, σε άλλες χώρες λαμβάνουν χώρα ετησίως. Δεν μπορεί λοιπόν ο καταναλωτής πιστεύω να θεωρεί ότι είναι ασφαλής γνωρίζοντας ότι σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στους ελέγχους. Η εναρμόνιση της συχνότητας των ελέγχων μπορεί να προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες διασφαλίσεις προστασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται κάποιες από τις τροπολογίες μου, με τις οποίες ζητώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει μέσω κατεξοδότηση υπράξεων ελάχιστες συχνότητες για κάθε προϊόν, διαδικασία ή δραστηριότητα. Ο κανονισμός θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει την διατροφική απάτη, στην οποία έχουμε εκτεθεί πολλά και στην Ευρώπη με το πρόσφατο σκάνδαλο, για παράδειγμα, του αλογιστικού κρέατος. Γι' αυτό θεωρώ ότι καλό θα ήταν να αναφέρουμε κέντρα αναφοράς, να εισάγουμε κέντρα αναφοράς ε, για την αυθεντικότητα και την ακαιρεότητα των ελέγχων των τροφίμων. Τηρώντας ταυτόχρονα τους κανόνες ευημερίας των ζώων ε, και ποιοτητα των τροφίμων. Για τα κράτη-μέλη που ε, χρησιμοποιούν τη δυνατότητα βαθμολόγηση των φορέων θα πρέπει να προβλέπεται κάποιο χρονοδιάγραμμα δημοσιοποίησης των πληροφοριών. Σε περίπτωση που ένας φορέας δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες, θα πρέπει να τον αγνωρίζεται η δυνατότητα, αφού έχει επανορθώσει η βαθμολόγησή του, η αξιολόγησή του να ενημερώνεται ταχύτερο δυνατόν. Τυχόν καθυστερήσεις θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες για τις δραστηριότητες. Από τα έγγραφα που έλαβα, ε, σχημάτισα την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια σύγχυση στην τερμηνία του κανονισμού. Γι' αυτό το λόγο ήθελα να διευκρινίσω ότι πέραν των γενικών κανονών για τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 8 της πρότασης κανονισμού ε, πρέπει να εφαρμοστούν και οι τομεακές. Από τα άρθρα 8 έως 14 έχουμε τους γενικούς κανόνες και από το 15 έως το 25 τους τομεακούς κανόνες. Τελευταία θα αναφερθώ στις εξαιρέσεις των μικρών επιχειρήσεων από την καταβόλη του υποχρεωτικού τέλους. Ε, τη βλέπω θετικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εξαίρεση των επιχειρήσεων αυτών. Θεωρώ όμως ότι τα κριτήρια που αναφέρει είναι υπερβολικά ευρεία. Όταν αναφέρεται σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους και με τζίρο χαμηλότερο από 2 εκατομμύρια ευρώ, το όλο σύστημα ελέγχων θα γίνει μη βιώσιμο. Τα κράτη θα πρέπει να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες με το δικό τους προϋπολογισμό. Η εξαίρεση πρέπει αυστηρά να περιορίζεται στις μικροεπιχειρήσεις και εγώ προτείνω το κατόφλιο των 200.000 ευρώ κύκλο εργασιών αλλά αυτό είναι απλά μια πρόταση για να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε μια τελική λύση, στην καταλληλότερη τελική λύση. Και ο τομέας των πρώτων υλών πρέπει να εξαιρεθεί, αλλά και εδώ θα ήθελα να συζητήσουμε για να δούμε τι απόψη έχουν οι συνάδελφοι. Τέλος, φαντάζομαι ότι θα ακούσουμε και παρατηρήσει για τις κατεξοδότηση πράξη, αλλά ήθελα να πω ότι αυτές οι πράξεις θα αποτελέσουν το εργαλείο εφαρμογής των παραρτημάτων της συγκεκριμένης τομαϊκής νομοθεσίας που ούτως ή άλλως συνεχίζει να ισχύει. Τέλος, στην τροπολογία 48, παράγραφος 1α, υπάρχει ένα σφάλμα. Έχει, υπάρχει κάποια παραπομπή στην παράγραφο 2. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τις άλλες τροπολογίες για να αφήσω περιθώριο για τις παρεμβάσεις των συναδέλφων που σίγουρος είμαι ότι θα είναι επικοδομητικές. Ευχαριστώ Μάριο Πυρίλο. Ο Ρίχαρτ Ζέμπερ α, αντικαθιστά τον κύριο Σνέλχαρτ ο οποίος βέβαια γνωρίζει πολύ καλύτερα ε, τα θέματα αυτά αλλά έπρεπε να πάει στη Γενική Συνέλευση των Χωρών ΑΚΕ και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Αλλά θα σας, ενημερώσω, θα σας ενημερώσει μέσω εμού. Ετοίμασε ένα κείμενο που θα το τηρήσω σχεδόν λέξη προς λέξη και βλέπει κάποιες ε, αμφιβολίες σε σχέση με τον κανονισμό 882 του 2004 που θα αντικατασταθεί από καινούριο που τον συζητάμε τώρα και που θα είναι καλύτερος ε, κάποια σκάνδαλα στην τροφική αλυσίδα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ε, υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Ο κύριος Σνέλχαρτ εντοπίζει τα εξή βασικά προβλήματα. Πρώτον, πεδίο εφαρμογής θεωρεί ότι δεν χρειάζεται όλες οι διατάξεις για τους επίσημους ελέγχους να συνοψίζονται σε μία νομική πράξη γιατί οι επιμέρους ε, ε, διατάξεις εφαρμόζονται καλά και μπορούν να παραμείνουν στα επιμέ... στους επιμέρους τομείς οι ανάλογες διατάξεις. Τώρα, για το name and shame, την ε, ε, ευθεία ε, κατηγορία των επιχειρήσεων όταν υπάρχουν σκάνδαλα, αυτό είναι καλό ούτως ώστε κάποιες ε, ύποπτες ε, ή ε, εταιρείες ή επιχειρήσεις που αδικοπρατούν θα πρέπει να είναι γνωστές στο κοινό. Βέβαια, αν σπεύσουμε να κατονομάσουμε μια εταιρεία, αυτό μπορεί να βλάψει το κύρος της και να επιφέρει μεγάλη ζημία σε μια εταιρεία που μπορεί να μην αποδειχθεί στο τέλος υπέτεια. Γι' αυτό Θεωρεί ο κ. Νέλχαρτ ότι χρειάζεται σαφής ορισμός του πότε οι αρχές δημοσιεύουν ποιες πληροφορίες, κυρίως όταν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν επιχειρήσεις και προϊόντα. Ένας άλλος τομέας που δημιουργεί προβλήματα στην κοινοποίηση είναι η κοινοποίηση επιμέρους αποτελεσμάτων ελέγχων και συστημάτων, συστήματα ταξινόμησης στα πλαίσια του ΙΜΠΕΛ γιατί αυτό είναι ένα ενσταντανέ ενώ η διαφύλαξη της, ε, των, ε, της ποιότητας των τροφίμων αποτελεί μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Έχει νόημα λοιπόν να μιλήσουμε για μακρότερο χρονικό διάστημα επί των οποίων θα υποβάλλονται εκθέσεις και αυτό νομίζω ότι καλύπτει και τα αιτήματα των ε, οργανώσεων των καταναλωτών. Ο Μάριο Πυρίλο ανέφερε τις νομικές πράξεις που δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα σε εμάς στο Κοινοβούλιο γιατί περιλαμβάνουν ε, διατάξεις ε, που περιλαμβάνονται στο δευτερογενές δίκαιο και δεν έχουμε εμείς δικαίωμα συναπόφασης. Τι χρειάζεται ο ελεγκτής ως πληροφορίες για να κάνει τη δουλειά του. Ε, αυτό δεν αναφέρεται στο βασικό δίκαιο. Και έτσι έχουμε ένα πρόβλημα, δηλαδή οι φυστάμενοι κανονισμοί χωρίς τα παραρτήματά τους ε, δεν ε, έχουν συμπεριληφθεί. Θα έπρεπε να συμπεριληφθούν λοιπόν. Βέβαια σε όλα αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί να αποφαίνεται με ναι ή όχι θα πρέπει το Κοινοβούλιο με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, και τη νομοθετική διαδικασία να ε, ενισχυθεί και να μην αποδυναμωθεί ως προς τις αρμοδιότητές του. Τέταρτον, η προβληματική των τελών. Όπως ξέρετε, υπάρχουν διατάξεις για τη νέα ρύθμιση των τελών. Ε, ο κ. Σνέλχαρτ θεωρεί ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε και να επεκτείνουμε δηλαδή τα τέλη και σε άλλους τομείς, θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που χρηματοδοτείται από από τους φόρους ε, βέβαια, αλλά ε, επειδή πολλά κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτό δεν είναι πολιτικά εφικτό, μπορούμε να έχουμε τα τέλη. Επίσης θεωρεί ότι η συμμετοχή των μεγάλων τομέων της οικονομίας ε, είναι, ε, η συμμετοχή τους είναι σωστή, αλλά θα πρέπει οι μεγαλύτερες να συμμετέχουν περισσότερο. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη ε, στοιχεία ε, πολύ συγκεκριμένα για τον ε, καθορισμό των μεγάλων επιχειρήσεων ε, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την αγοραστική δύναμη των κρατών μελών. Θεωρεί ότι και αυτή, αυτό το, ο γραφειοκρατικός φόρτος θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και να βρεθεί κάποια ισορροπία. Ε, ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι είναι πάρα πολλές οι μικρομεσαίες στον τομέα των τροφίμων. Αυτό είναι το κείμενο του Χορ Σνέλχαρτ ε, θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στο θέμα των τελών που είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα όταν οι εταιρείε τροφίμων πληρώνουν τους ελεγκτές οι ίδιες ε, εκεί είναι ευαίσθητο το θέμα και πρέπει να προσέξουμε για να μην το παρακάνουμε και η αρχή name and shame είναι σημαντική. Ζούμε σε μια κοινωνία των μέσων, των ενημέρωσης. Ε, και ε, είναι πολύ επικίνδυνη η κριτική, ιδιαίτερα όταν από επίσημες πλευρές δεν είναι βέβαιες, βέβαιες οι κατηγορίες. Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί ελέγχων που παρεμβαίνουν και ε, καλύπτουν ε, όλον αυτό το τομέα και την κοινοποίηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος... Όχι, η κυρία Πάουλσεν δεν είναι εδώ. Ο Μπερτ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρετίζω την έκθεση Πυρίλο. Θα πρέπει να εξετάσουμε το γενικό πλαίσιο καταρχήν όλα τα ε, διατροφικά σκάνδαλα υποσκάπτουν την ε, εμπιστοσύνη του καταναλωτή οπότε ε, χρειάζεται η έλεγχη να είναι αυστηρή έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Για τη δική μας πολιτική ομάδα ο κανόνας, ε, ο βασικός κανόνας θα πρέπει να είναι ότι οι, εθνικές, αρχές θα πρέπει να διενεργούν επαρκή αριθμό ελέγχων, θα πρέπει να μεριμνούν έτσι ώστε να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, επαρκές προσωπικό, τα επαρκή μέσα και το προσωπικό θα πρέπει να ε, έχει επιμορφωθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Όλα αυτά είναι προφανή, αλλά στην πραγματικότητα ε, τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Την περασμένη εβδομάδα στη χώρα μου, το Βέλγιο, ε, μια επιθεώρηση απεκάλυψε ότι οι εθνικές μας αρχές ελέγχου που παλιότερα ήταν ε, ε, πολύ ικανές ε, χρειάζεται ε, χρειάστηκε εξαιτία των μέτρων λιτότητας να κάνει περικοπές και η μείωση του προσωπικού των μέσων που διαθέτει οδηγεί σε μείωση της, οδήγησε σε μείωση της αποτελεσματικότητάς της. Χρειάζεται επίσης μια στενή συνεργασία ανάμεσα στις αρχές ελέγχου το σύστημα επαγρύπνησης λειτουργεί πολύ, πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Ε, θα υπερψηφίσουμε και την έκθεση για την απάτη στον αγροδιατροφικό, αγροτροφημικό τομέα. Χρειάζεται ένα σύστημα επαγρύπνησης και σε μας ε, γιατί ε, αυτό δεν έχει σχέση τόσο με τη δημοσιακή υγεία όσο με την προστασία των καταναλωτών. Είναι δυνατόν να φανταστούμε και συστήματα αυτοελέγχου, αλλά νομίζω ότι η επίσημη έλεγχη από τις εθνικές αρχές θα πρέπει να είναι αποφασιστική σημασία. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι αρχές ελέγχου θα πρέπει να αναλύουν ε, τον κίνδυνο και να γίνονται και ξαφνικές ε, ε, ευνηδιαστικές συγγνώμη επιθεωρήσεις Ε, <clears throat> όχι μόνο βέβαια ευθυνδιαστικές ε, ε, επιθεωρήσεις, θα πρέπει να υπάρχουν και προγράμματα επιθεωρήσεων, αλλά ε, θα πρέπει να γίνονται και ευθυνδιαστικές επιθεωρήσεις. σε ό,τι διάφορα τους τους σε ό,τι αφορά το, το ακαθόδες θέμα του, της χρηματοδότησης, να πω το εξής. Η, όλες οι αρχές υφίστανται πιέσεις, ε, οικονομικές πιέσεις, πρέπει να ε, μειώσουν τον προπολογισμό τους. Ε, θα πρέπει όμως να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στους ελεγχόμενους και τους ελεγκτές. Δηλαδή μπορούν και οι ελεγχόμενοι να συμμετέχουν κατά κάποιο τρόπο στους ελέγχους με αυτοέλεγχο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στους δύο. Η ε, αρχές ελέγχου θα πρέπει επίσης να είναι ανεξάρτητες. Θα πρέπει να προέρχονται από το Υπουργείο ε, Υγείας και όχι από το Υπουργείο Γεωργίας. Όταν έγινε η Ειδική Επιτροπή για την ως των τρελών αγελάδων, ε, μεταφέραμε την αρμοδιότητα με την Επιτροπή Γεωργίας στην Επιτροπή Δημόσιας Υγείας. Βλέπω όμως ότι σιγά σιγά το Υπουργείο Γερία στη χώρα μου ε, έχει ξαναπάρει το πάνω χέρι. Ε, αυτό όμως δεν είναι σωστό. Σε ό,τι αφορά την διαφάνεια, είμαι υπέρ της μέγιστης δυνατής διαφάνειας. Θα πρέπει να δημοσιεύονται βέβαια γεγονότα, ε, στοιχεία τα οποία να είναι αξιόπιστα, ενώ η διαφάνεια θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να αποδεικνύεται και η ποιότητα των ελέγχων που διενεργούνται. Επιπλέον, είναι καλό να τα ελέγχουμε όλα βέβαια, αλλά θα πρέπει να επιβάλλουμε και αρκετές κυρώσεις. Και μάλιστα κυρώσεις οι οποίες να είναι παρκώς αυστηρές. Αν οι κυρώσεις που επιβάλλονται δεν είναι αρκετά αυστηρές, δεν θα έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο αποθαρρύνονται οι ίδιοι επιθεωρητές. Αυτές είναι οι ιδέες της ομάδας μου και με βάση αυτές θα υποβάλουμε τροπολογίες. Ευχαριστώ. ECR, παρακαλώ. Julie ECR. Thank you. Um, I'll be... Ευχαριστώ πολύ, θα είμαι σύντομη. Ευχαριστούμε τον κύριο Περίλο για την εκθεσή του. Η κυρία Γκέρλινγκ. Αυτό που διακρίνω εγώ σε όλη την έκθεση είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για την επικουρικότητα. Σε πολλούς ε, τομείς ε, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ε, ότι τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνες και πρέπει να προσέξουμε να μην θολώσουμε αυτά τα αέρια. Με ανησυχεί η έκταση και η ποσότητα των κατεξουδότηση πράξεων. Υποτίθεται ότι μειώνουμε το διοικητικό φόρτο. Υποτίθεται ότι προχωράμε σε απλούστευση. Αλλά με πολλούς από αυτούς τους κανονισμού πλαίσια τελικά αναρωτιόμαστε μήπω τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, πιο περίπλοκα. Μήπως είναι πιο περίπλοκο να δει κανεί ποιο είναι υπεύθυνο γιατί, ποιο είναι αρμόδιος γιατί. Είναι πολλά τα άρθρα και κάθε σημείο πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά. Οι χρεώσεις που αναφέρονται δεν λαμβάνουν υπόψη τις διεθνότητες του κάθε κράτους μέλους και τις ε, όρους πρακτικής εφαρμογής. Ε, νομίζω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν την ευθύνη να αποφασίσουν εδώ και να αναλάβουν το καθήκον, να διασφαλίσουν ότι ε, θα εγκατασταθούν επαρκείς έλεγχοι σύμφωνα με το πλαίσιο. Και η χρέωση θα πρέπει να γίνεται σωστά. Δεν λέω πώς πρέπει να καταβάλλονται οι πληρωμές, γιατί κάτι τέτοιο θα δυσχέρανε την κατάσταση. Καλωσορίζω την τροπολογία 39 του κυρίου Πυρηλό όσον αφορά τους ε, πρωτεύοντες παραγωγούς. Εγώ εργάστηκα στους οριζόντους κανονισμούς της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής και γνωρίζω ήδη ότι μέσω της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, συμβάλλουν οι αγρότες στις επιθεωρήσεις και δεν χρειάζεται να πληρώνουν. Αυτό θα επηρεάσει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και όλοι οι φορείς ε, μετακυλίουν το κόστος ε, στο πρώτο παραγωγό χωρί την τροπολογία του κυρίου Περίλου. Θα σας έλεγα λοιπόν να το ε, εξετάσετε προσεκτικά. Οι πρωτογενείς παραγωγοί δεν έχουν να μετακυλήσουν το κόστος σε κανέναν. Ενώ υφίστανται ταυτόχρονα πολύ μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή όσον αφορά την κερδοφορία. Και ξέρετε, αν ένα αγρόκτημα δεν είναι επικερδές, δεν είναι και βιώσιμο και πρέπει να φροντίσουμε να μην επιβάλλουμε περισσότερο φόρτο σε αυτή την κατηγορία. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για τα τρόφιμα. Φυσικά αυτή η επίσημη έλεγχη που προτείνονται προτείνονται λίγο μετά τα προβλήματα με το λογισιο κρέας και συνάδουμε τη δική μας έκθεση πρωτοβουλίας πρέπει είναι σημαντικό να μην συγχαίρουμε και ποια ζητήματα εδώ. Υπάρχει διαφορά μεταξύ επίσημων ελέγχων και ελέγχων των τροφίμων. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το θέμα εδώ. δεν πρόκειται απαραίτητα να αποτελέσει μέσο ελέγχου των τροφίμων. Φυσικά αποτελεί βάση, ένα πλαίσιο, ώστε να γνωρίζουμε κατά πόσο οι επιχειρήσεις ε, της ελισίδας έχουν κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουν, αλλά εν τέλει η, ο εντοπισμός των ε, απατών ε, θα βασιστεί σε μηχανισμούς ε, εντοπισμού, επιτόπου ελέγχους, δηλαδή θα βασιστεί στο ότι ο κόσμος δεν θα γνωρίζει πότε θα ελεγχθεί σε ολόκληρη την αλυσίδα. Φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε υπερβολικά αυστηρού κανόνε γιατί θα μάθουν ποιοι είναι οι κανόνε. Αλλά πρέπει να έχουμε ένα ευέλικτο σύστημα ώστε να είναι αυτή η ελέγχη δυνατή η απρόβλεπτη ελέγχη και ίσω η νομοθεσία αυτή να μην είναι το καλύτερο σημείο να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή αποτελεί απλά μια βάση. Thank you very much. Κρίστοφα Φιέλνερ και μετά η Λίντα Μακαϊβάν. Ευχαριστώ. Αν μου ε, είχε πει κανείς ε, πριν από δύο εβδομάδες αν ήθελα να συζητήσω το θέμα, θα έλεγα μάλλον όχι. Πριν καταλάβω ότι εδώ ε, ελέγχουμε τα πάντα και είναι ευρύτατος ο κανονισμός αυτός για τους ελέγχους, το θέμα που με έκανε να θέλω να συμμετάσχω στη συζήτηση και κατέθεσα και τροπολογίες μάλιστα είναι ότι κατάλαβα ότι τώρα με αυτόν τον κανονισμό έχουμε κοινό κανονισμό για το αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτά που πάνε για ανθρώπινη κατανάλωση. Όλα αυτά θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται και πολλές φορές με διαφοροποίησεις. Καλό θα ήταν να υπάρξει η να συνεχιστεί να ισχύει η φυστάμενη οδηγία. Γιατί? Γιατί δεν έχει πρόβλημα. Γιατί να το διορθώσουμε, να διορθώσουμε. Προετοιμαζόμενος μίλησα με εκπροσώπους πολλών κρατών μελών, μίλησα και ε, είδα και το υλικό που είναι η βάση του κανονισμού και όταν εξέτασα το υλικό μας κατάλαβα ότι όλα τα κράτη-μέλη ήθελαν λίγο πολύ να διατηρήσουν την υφισταμένη οδηγία για το υλικό αυτό και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε ε, αν ε, άλλαζε να δημιουργήσει ε, πρόσθετο φόρτο σε όλους. Αν πρόκειται να εφαρμόσουν τους ίδιους κανόνους για το υλικό που προτίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Δεν χρειάζεται λοιπόν διόρθωση για τον απλούστατο λόγο ότι η οδηγία είναι και σχετικά καινούρια, είναι του 1999 και μία από τις λίγες οδηγίες που εφαρμόστηκαν ε, πολύ καλά από όλα τα κράτη-μέλη. Επειδή λοιπόν είναι μόνο ηλικίας 10 ετών, είναι σχετικά ενημερωμένες οι διατάξεις που περιέχει και δεν βλέπω λόγο να ενημερωθούν ξανά οι διατάξεις στα πλαίσια αυτού του κανονισμού. Όμως, αν επιλέγαμε την ε, πρόταση της Κομισιόν, για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά με τον ίδιο τρόπο, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το ε, ε, ε, θα είχαμε αυξημένες δαπάνες για τη διαχείριση. Γιατί αν είχαμε το ίδιο σύστημα συμμόρφωσης ή χνηλασιμότητας που προβλέπετε εδώ, δεν θα με εξέπλητε αν κάποιοι ιδιοκτήτες θα ήθελαν να μειώσουν την ποικιλότητα. Ε, για να ανταποκριθούν στα, στις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. Ή όταν μιλάμε για φυτά, για ανθρώπινη κατανάλωση, εκεί βέβαια η ιχνηλασιμότητα έχει μεγαλύτερο η ηχνηλασιμοτητα εχει Αλλά δεν έχει όταν μιλάμε για τα δασικά προϊόντα και τη δασοκομεία. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι σίγουρα χρειάζεται μια γενική ενημέρωση, οριζόντια και η θέσπιση του κανονισμού, αλλά πρέπει να εξετάσουμε ιδιαίτερα κάποιες λεπτομέρειες. Γι' αυτό εγώ επικεντρώθηκα στα δασικά, γιατί το ξέρω το θέμα. Υπάρχουν όμως και άλλοι τομείς ενδεχομένως που αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, ενώ δεν θα έπρεπε αναγκαστικά. Αυτό άλλοι θα το κρίνουν. Πάντως πρέπει να αξιολογήσουμε όλες τις πτυχές, όλα τα βήματά μας ένα προς ένα. Τουλάχιστον όμως ε, να πούμε ότι το αναπαραγωγικό δασικό υλικό θα πρέπει να μείνει απ' έξω και να ισχύσει η φυστάμενη οδηγία. Η Λίντα Μακαϊβαν και μετά η Πιλάρα Γιούζο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Σίγητη που ανέλαβε ένα τέτοιο περίπλοκο θέμα. Κρίμα που γίνεται αυτή η συζήτηση στο Κοινοβούλιο τόσο αργά στη θητεία του Κοινοβουλίου αυτού. Τόσα πολλά νομοθετήματα φτάνουν σε τελική φάση και φοβάμαι ότι δεν θα πρόλαβουμε να εξετάσουμε αυτό το τεράστιο νομοθέτημα που συγκεντρώνει τόσο πολλές νομοθετικές πράξεις. Ανησυχώ για αυτούς τους ε, μέγα νόμους που προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα πάντα και για το πλήθος των κατεξιδότηση πράξεων που δημιουργούνται από τέτοια νομοθετήματα. Η εμπειρία με κάποιες κατεξιδότηση πράξεις στον τομέα των τροφίμων ε, δεν με καθησυχάζει ιδιαίτερα. Δεν ξέρω κατά πόσο οι αποφάσει πρέπει να λαμβάνονται από τεχνικές επιτροπές, γιατί οι αξιωματούχοι συχνά δεν θέλουν να λάβουν ε, μη δημοφιλείς αποφάσεις, δυσάρεστες αποφάσεις, οπότε δεν λαμβάνουν καμία απόφαση και πρέπει να εξετάσουμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το πλήθος των τη πράξεων εδώ. Ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν. Ξέρω ότι πολλά χρόνια έχει διαρκέσει η εκπόνηση αυτού του νόμου. Όταν συζητήσαμε εδώ με τον Γενικό σας Διευθυντή και τον Επιτρόπο, μας είπαν ότι αποκομίστηκαν διδάγματα και έχουν ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ποια διδάγματα αποκομίσατε και ενσωματώσετε σε αυτήν εδώ την νομοθεσία. Διότι αυτή είναι μια ευκαιρία να τα εντάξετε εδώ τα διδάγματα που αποκομίσατε. Κάποια θέματα αναφέρθηκαν από του συναδέλφου, η ανεξαρτησία των ελέγχων, ειδικότερα στην επιθεώρηση των κρεάτων. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στα σφαγεία δεν κάνουν και την ευκολότερη δουλειά του κόσμου. Δεν είναι ένα μέρο που μπορεί κάποιο να πάει στο αφεντικό και να πει: Κοίτα, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Μπορεί να ρίξει μια ματιά. Διότι κινείται γρήγορα η δραστηριότητα και οι συνθήκες εργασίας δεν είναι και οι καλύτερες για πολύ κόσμο και η δυνατότητα ορισμένων εργαζομένων να αμφισβητήσουν τη διοίκηση δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλη. Τι σημαίνει ακριβώς λοιπόν εξυγχρονισμός. Διότι μιλάμε για εξυγχρονισμό εδώ και χρόνια και παλιά εννοούσαμε απελευθέρωση, λιγότερους κανονισμούς για το καθεστώς ελέγχου των κρέατων. Κάτι που προέκυψε μετά από το σκάνδαλο του αλογίσιου κρέατος ε, αφορούσε τον συχνότητα των ελέγχων. Τα, οι εγκαταστάσεις κοπής ε, που είχαν πιο συχνές ε, επιθεωρήσεις και σήμερα δεν επιθεωρούνται καθόλου. Τι γίνεται με αυτό. Όταν μίλησα με κάποιον υπεύθυνο στην Αγγλία για την επιθεώρηση των κρεάτων μου είπε ότι κάποια βιομηχανίες ε, ελέγχονται πολύ διότι κάποιο σούπερ μάρκετ στέλνουν τους δικούς επιθεωρητές. Ορισμένα δηλαδή οι σφαγεία ελέγχονται και από δικούς τους ελεγκτούς, ελεγκτές. Ε. Ορισμένες όμως εγκαταστάσεις αλλά κάποιες μικρές εγκαταστάσεις αυτό δεν συμβαίνει. Δεν μπορούμε λοιπόν να βασιστούμε στο γεγονό ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ επιθεωρούν ορισμένε εγκαταστάσει. <coughs> Αυτό δεν μα καθησυχάζει ότι είναι ασφαλή και τα κράτα βγαίνουν από μικρότερες εγκαταστάσει. Δεν θέλω να μα το σχολιάσει αυτό η Κομισιόν. Υπάρχει πια διάταξη γι' αυτό. Και τι γίνεται στι εγκαταστάσει Κοπή. όσον αφορά τι επιθεωρήσει, όχι μόνο στη σφαγεία. Και τέλος, ε, η ορολογία που συζητείτε εδώ είναι ασφάλεια τροφίμων. Τις προάλλες συζητήσαμε τις αλλαγές της επιθεωρής των κρεάτων. Ακούσαμε να μιλάει ο κόσμος για ποιότητα των τροφίμων. Για τις δυνατότητες, τις πιθανότητες ε, ε, να υπάρξουν προϊόντα που ο κόσμος μπορεί να μην θέλει να φάει, να μην θέλει να περιέρχονται στα τρόφιμα που τρώει. Όχι απαραίτητα που θα οδηγήσουν σε ασθένειες. Θέλω λοιπόν να μου μιλήσουμε για την καθαρότητα των τροφίμων, για το πόσο σωστά είναι. Μιλάω για τις περιπτώσεις τις οποίες χρησιμοποιούνται που χρησιμοποιούνται μείγματα διαφόρων ε, κρεάτων. Δεν υπήρχε κάποια διάταξη για την επισήμανση των τροφίμων. Ο κόσμος όμως ανησυχεί για την ποιότητα, για την καθαρότητα των τροφίμων. Φοβάμαι ότι κοιτάτε την ασφάλεια των τροφίμων μόνο, αλλά δεν καλύπτει αυτό το ζήτημα. Πώ μπορεί να γνωρίζει το κοινό τι ακριβώ τρώει. Ευχαριστώ. και μετά η κυρία Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή κύριο Πυρίλο τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα. Σε γενικές γραμμές, ε, συμφωνώ με τον κύριο Έσνερ, Έχω όμω να κάνω τα εξή σχόλια. Έχουμε κάποιε αμφιβολίε για το κατά πόσο πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο του κανονισμού σε όλου του τομεί. Συμπεριλαμβανομένου και των δασοκομικών ε, φυτών και των ε, σπόρων σε φυτόρια που δεν αποτελούν τμήμα της διατροφικής αλυσίδας. Επίσης θα πρέπει να διευκρινίσουμε αν η οικολογική παραγωγή ε, γεωγραφικών ενδείξεων και προελεύσεων και ε, ονομασιών προέλευσης συμπεριλαμβάνονται ή όχι. Επίσης πρέπει να διευκρινίσουμε τους, ελέγχους, τους ε, ορισμούς των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων ελέγχων, γιατί στην σημερινή διατύπωση του κειμένου δεν υπάρχει σαφήνεια. Ίσως θα πρέπει να διαγράψουμε το κεφάλαιο των άλλων επίσημων ελέγχων. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι έλεγχοι είναι επίσημοι. Εν πάση περιπτώσει η πρόταση κάνει διάκριση ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη. Η Επιτροπή προτείνει πολλές ε, πράξεις κατά εξουδότηση και εκτελεστικές πράξεις ενώ υπάρχουν και διατάξεις για επίσημους ελέγχους των κρατών μελών, τα, οι οποίοι δεν θα πρέπει να είναι ε, αρμοδιότητα της Επιτροπής. Όσο οι, τα κράτη-μέλη σέβονται τους, τους κάθε κρατός θα πρέπει να μπορεί να ε, οργανώνεται όπως θεωρεί απαραίτητο. Μετά, σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των ελέγχων, η Κομισιόν προτείνει ε, τα τέλη που θα εισπράττονται να τα διαχειρίζονται οι υγειονομικές ε, αρχές για τη χρηματοδότηση των ελέγχων. Όμως υπάρχουν φορολογικά στήματα σε διάφορα κράτη-μέλη, όπως η Ισπανία για παράδειγμα, που η, το Υπουργείο Οικονομικών ε, συλλέγει και αναδιανέμει αργότερα αυτά τα τέλη. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό σε μια τροπολογία. Μετά, έλεγχη εξαγωγών. Αυτό, αυτοί αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οπότε η ε, Κομισιόν δεν είναι δυνατόν να αναλάβει αρμοδιότητα σε αυτό το τομέα. Είναι θέμα διμερών συμφωνιών μεταξύ της χώρας που εξάγει και της χώρας που εισάγει. Ε, μετά, η Κομισιόν θέλει επίσης να παρέμβει και στις επιθεωρήσεις σε τρίτες χώρες, μάλλον και σε επιθεωρήσεις που ε, τρίτες χώρες κάνουν στα κράτη-μέλη πριν ε, δώσουν την άδεια για εξαγωγή. Και εδώ νομίζω ότι η Κομισιόν ξεφεύγει των αρμοδιοτήτων της, είναι θέμα διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Η Ντάκμα Μπέρεν και μετά ο Τζον Στιουαρτ. Μισό λεπτό. Υπάρχει άλλος ομιλητής πριν. Προηγείται άλλος. Η Ντάγμαρ. Ευχαριστώ Ματίας. Έχω μια αίσθηση déjà vu ακούγοντας αυτές τις συζητήσεις. Δίσταζα να ζητήσω το λόγο. Γιατί ειλικρινώς καμιά φορά πιστεύω ότι καλύτερα είναι να μην μιλάει κανείς. ενώπιον ανθρώπων που μα ξέρουν καλά και για πολύ, εδώ και πολύ καιρό. Εκτός από τον Μπέρτ Στάις και εγώ όμως, λίγοι ξέρουν τόσα πολλά τα τρόφιμα, τους ελέγχους και τους λόγους για τα σκάνδαλα. Ακούγοντας ορισμένους από εσά και την συνάδελφο Γκέρλινγκ που δυστυχώς έπρεπε να φύγει, βλέπω ότι είναι από άλλο κόσμο λένε ότι είναι σημαντικό να τηρήσουμε την επικουρικότητα και ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να το χειριστούν σωστά. Τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό είχαμε το σκάνδαλο με τη σφουγγόδια εγκεφαλοπάθεια. Επειδή ήταν τα κράτη-μέλη αποφασίσαμε να μην υπάρχει επισήμανση ε, για ε, τρόφιμικες ζωοτροφές, ε, για φυτοφάγους από όταν είχαμε προϊόντα από ζωά αγελάδες. Τα κράτη-μέλη έπρεπε να αποφασίσουν ότι ήταν δυνατόν να έχουν φτηνές ζωοτροφές ε, και τα κράτη-μέλη αφού διαπίστωσαν ότι υπάρχει σκάνδαλο με μολυσμένα ζώα και ότι θα υπήρχε η δυνατότητα, η πιθανότητα και οι άνθρωποι να προσβληθούν και να πάθουν όχι την ασθένεια των ζώων αλλά την ανθρώπινη εκδοχή που ήταν η Κρόιτσφελτ Γιάκομπς. ναι, τα κράτη-μέλη ε, είχαν την αρμοδιότητα και τα έκαναν όλα αυτά. Και ποιος θα δείξει εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη ότι ενδιαφέρονται για τους ελέγχους. Βέβαια, παίζει ρόλο ο χαρακτήρας του καθενός, αλλά η κατάσταση δεν είναι ρεαλιστική. Και ε, εκτιμώ αυτό που έκανε ο Μάριο Πυρίλο. Δούλεψε σκληρά. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με την τροπολογία 39, γιατί εκεί μου φαίνεται ότι είμαστε κάπως υπεραισιόδοξοι που ε, εμπιστευόμαστε τους παραγωγούς επιτόπους και την προπαραγωγή. Εκεί έχω κάποιες αμφιβολίες, είναι το μόνο σημείο. Όμως Θέλω να νερώσω λίγο αυτό το κρασί του ενθουσιασμού μας. Όταν μιλάμε για ελέγχους και πραγματικά ε, ακούσαμε ε, και υπεύθυνε απόψεις εδώ, ε, εδώ αντλήσαμε μαθήματα, διδάγματα και τα κράτη-μέλη επίσης. Μπορούμε να νομοθετήσουμε άψογα εδώ και ελπίζω ότι θα είναι σχεδόν τέλειο το νομοθέτημά μας όταν τελειώσουμε. Αλλά αμφιβάλλω αν, ε, ακούγοντας ορισμένους όπως τη συνάδελφο Γκέρλινγκ που πρέπει να ε, πείσει την κοινή γνώμη ότι δεν προτίθενται να κάνουν τέλειους ελέγχους και ότι θέτουν σε κίνδυνο τους καταναλωτές. Ας το αναλάβει εκείνη. Εκείνοι ε, που έχουν αυτές τις απόψεις βάζουν σε κίνδυνο τους καταναλωτές. Ε, εμείς ε, είμαστε ένα σώμα 28 κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πολλά εκατομμύρια κατοίκους. Δεν μπορεί να έχουμε ένα εκατομμύριο ελεγκτές. Πάλι λοιπόν ε, ε, βασιζόμαστε στην αποτελεσματικότητα των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη θα μας παρασταθούν, θα είναι διατεθειμένα να επενδύσουν σε, περισσότερες και, σε περισσότερους και καλύτερους ελέγχους. Όχι. Δείτε το τελευταίο νομοθέτημα που εξετάσαμε για τους ε, ελέγχους τους χείρους, τα σφαγεία. Δεν ξέρω αν έχετε, πόσοι από εσά έχετε πάει πρωί στο σφαγείο που δουλεύουν ή αν έχετε πάει σε ένα ε, μια μονάδα αδρανοποίησης ε, ε, σε ένα τεμαχιστήριο. Να πάτε, πηγαίνετε σε τεμαχιστήριο. Εγώ έχω πάει και ξέρω τι κλίμα επικρατεί, ξέρω την ταχύτητα με την οποία δουλεύουν. Είναι αυταπάτη αυτό που κάνουμε αν αποδυναμώσουμε τις διατάξεις για όλα αυτά ε, και βεβαίως ε, ε, εκτιμώ τους ανθρώπους από την DG Sanko που ετοίμασαν την κατεξουσιοδότηση πράξη και προτείνουν την μείωση των ελέγχων στους χείρους δηλαδή να είναι μόνο έλεγχη εποπτείας και όχι στο δημαχιστήριο. Ε, όμως δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε όλες τις διατάξεις που έχουμε. Ε, να συνεχίσω με βάση αυτό που είπε η Λίντα, αλλά βέβαια από την Κομισιόν θα μπορούσατε, δεν θα μπορούσατε, αλλά προσπαθήστε να μας πείτε τι διδάγματα αντλήσατε και πού υπάρχουν αυτά στις προτάσεις και τι λένε τα κράτη-μέλη. Αυξάνουν τους ελέγχους. Την απάντηση την ξέρουμε και οι δύο. Ε, θέλουμε να διευκρινίσουμε το θέμα. Θυμάστε ε, όταν θέλαμε την επισήμανση για την χώρα προέλευσης για το επανεπεξεργασμένο κρέας. Το καταφέραμε. Ε, είχε γίνει στην Κομισιόν ε, αν, εκτίμηση αντικτύπου. Είναι, ξέρω, ξέρω, είναι, είναι τα τελευταία 15 χρόνια το θέμα που χειρίζομαι. Ξέρουμε ότι γίνεται έλεγχος επιπτώσεων είναι πάρα πολύ δαπανηρό και οι καταναλωτές δεν θέλουν προ... τη χώρα προέλευσης. Αυτό ε, είπατε. Ποιος όμως θα αποφάσισε αυτό ότι δεν θέλανε. Ας γίνει μια έρευνα τώρα πριν από τις ευρωεκλογές. Το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό από αυτό που έχει μπροστά τη η Κομισιόν. Η έκθεση είναι καλή. Ο Μάριο Περίλο έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει εκτό από την τροπολογία 39. Αλλά ε, ε, τώρα τα κράτη-μέλη είναι ε, αρμόδια και ε, ε, τα κράτη-μέλη δεν θα επενδύσουν, ε, δεν θα κάνουν περισσότερους ελέγχους, δεν θέλουν καλύτερο σύστημα από αυτό που είναι τώρα, οπότε διατρέχουν κίνδυνο οι καταναλωτές. Θέλουν να αποδυναμώσουν τις διατάξεις και όχι να τις ενισχύσουν. Μάλιστα. Τώρα τελείως, όχι, ο Τζον Στιούαρτ Άγνιος. Συγγνώμη που προσπάθησα να υπερκεράσω το, την να μιλήτρα για να πάρω τη σειρά τη, αλλά ήταν πολύ ωραίο που την άκουσα. Θέλετε να με ακούσετε παρακαλώ. Γιατί ε, ισχυρίζεστε ότι ξέρετε πολύ περισσότερα για τι ασθένειε των ζώων και τη μεταχείριση των ζώων από μένα. Εγώ είμαι γεωργός, είμαι κτηνοτρόφος. 600 ε, προβατίνες χρειάστηκε εγώ να δω να πεθαίνουν ε, γιατί τις φάξανε ε, ε, για να μην μεταδοθεί ασθένεια χωρίς να έχουν τίποτα. Ε, ούτε καν μας ασφαλίζουν γιατί φοβούνται τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ε, αν είχαμε ένα θετικό δείγμα σαλμονέλας, τι θα γινόταν, αυτό να ρωτιόμασταν. Ε, Όμω είναι τόσο αποτελεσματικό το σύστημά μα που όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Οπότε οι ασφαλιστικέ εταιρείε άρχισαν να μα ασφαλίζουν. Που, από πού ήρθε το πρόβλημα τη Αλμονέλα. Από εισαγμένα ισπανικά αυγά, δεν είχε σχέση με εμά. Μετά είχαμε την, ενός, τη, τη των πτηνών. Μετά έπεσαν στο κεφάλι μας όλοι οι κανονισμοί. Εμένα με επιθεωρούν σχεδόν κάθε εβδομάδα από ε, ο, α ή ο β φορέας, δεν έχει σημασία ποιος. Έχω πάρει χιλιάδες ε, mail για αυτό το θέμα. Ποιοι διαμαρτύρονται για τον Πυρίλ, για τον Πυρίλ δεν ε, μιλάμε. για τον απαραγωγικό υλικό. εδώ συνδέονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένα κόμμα μόνο ανάμεσά τους. Τι, δεν έχω τη σωστή ημερήσια διάταξη. Το 4. Κανόνε για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό. Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, Πρόεδρε. Στη μέση διάταξη είναι. Okay, vielen Dank. Die britische Kuh wird ja... Ευχαριστώ. Οι βρετανικές ε, αγελάδες ε, εξετάζονται από πολλούς ε, διαφορετικούς φορείς, όχι όμως οι Βρετανοί αγρότες. Αυτό σύμφωνα με μια έρευνα. Η Κορίν όχι, επιβεβαιώνω ότι μπορώ να μιλήσω για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που το λέει και η μερίσια διάταξη. Δεν μπορώ να λάβω το λόγο επ' αυτού. Είμαστε στο σημείο 4, όχι στο σημείο 7. Αυτό που λέτε είναι για το 7. Ευχαριστώ η Κορίν Λεπάζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συντομία ήθελα να συμφωνήσω με τα όσα είπε η κυρία Ροτμπερέντ ε, και ο κύριος Στάς. Είναι ένα θέμα για το οποίο εμείς οι ευρωβουλευτές έχουμε δίτρη ευθύνη. Μιλάμε για θέματα για τα οποία έχουν προσδοκίες από εμάς οι πολίτες μας ε, ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στο ότι καταναλώνουν γενικότερα. Ε, Αν ναι, εμείς ε, δεν είμαστε ιδιαίτερα απαιτητικοί για όλα τα συστήματα και για τους πραγματικούς ελέγχους, δεν εκπληρώνουμε την αποστολή μας. Δεν πρέπει λοιπόν να διστάσουμε σε αυτά τα σημεία. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι έχω σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά το πλήθος των κατεξιοδότηση πράξεων που προβλέπει το κείμενο αυτό. είναι σαν να ρίχνουμε τις ευθύνες μας ε, στην Κομισιόν. Δεν είναι αποδεκτό σε τόσο μεγάλο βαθμό. Thank you, uh, Mrs. Lepage. Ευχαριστούμε κυρία Λεπάζ. Ήταν η τελευταία ομιλήτρια από πλευρά Κοινοβουλίου. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω την κυρία Κέρμαν Καρό. Το είπα σωστά. Uh, thank you. That is correct, Mr. President. Um, thank you. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον εισηγητή. Είναι πολύ επικοδομητική η έκθεσή του. Οι ιδέες του γενικά ε, έχουν ως στόχο τη βελτίωση πρόταση κομισιών. Θα κάνω μερικά σχόλια και μετά θα απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Σε ό,τι φορά τα τέλη και τις εξαιρέσεις από την πληρωμή των υποχρεωτικών τελών για μικρόμεσες επιχειρήσεις. Να σας υπενθυμίσω τη λογική πίσω από την πρότασή μας. Ε, η λογική είναι ότι θέλουμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη, ε, στις αρχές των κρατών μελών, τους απαραίτητους πόρους, προκειμένου να παίξουν το ρόλο τους, να συνεχίσουν δηλαδή να διατηρήσουν ένα αποτελεσματικό επίπεδο ελέγχων Από εκεί, γι' αυτό ήταν σημείο αφετηρία τη Κομισιόν, ότι δηλαδή οι, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και οι περικοπέ οδηγούν στη μείωση των επίσημων ελέγχων και ενδεχομένως πια δεν είναι επαρκή για το επίπεδο κινδύνου το οποίο εντοπίζεται στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Σκεφτείτε το αυτό, έχετε το στο μυαλό σα, διότι εξαιρώντας τις πιο ευαίσθητες ευάλωτες επιχειρήσεις, οι εξαιρέσεις αυτές δεν σωρεύονται έτσι ώστε το σύστημα να γίνει μη βιώσιμο. Τι εννοώ. Εννοώ ότι το σύστημα είναι περίπλοκο το εννοώ ε, το, σύστημα για τον υπολογισμό του κόστους των τελών, τη σύσπραξη των τελών κλπ. Η, αλήθεια είναι ότι είναι σημαντική προσπάθεια που απαιτείται από τα κράτη-μέλη. Και επειδή ακριβώς είναι σημαντική θα πρέπει να αξίζει τον κόπο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα περίπλοκο σύστημα για να εισπράττουμε ένα πολύ μικρό ποσό σε σχέση με το αναγκαίο για να γίνονται οι έλεγχοι. Τώρα σε ό,τι αφορά τις ε, ε, ε, ε Δεδομένου ότι καταργούμε κάποιες ε, διατάξεις και ενοποιούμε κάποιες άλλες, χρειάζονται οι καταξιδότηση πράξεις ε, και μάλιστα τις ε, ε, ομαδοποιούμε. Δεν θέλουμε με αυτές τις πράξεις να αλλάξουμε τη σημερινή κατάσταση. Οι εξουσίες τις οποίες ζητάει η Κομισιόν θα επιτρέψουν να, μας, ε, να, να συνεχίσουμε να νομοθετούμε για τις ανάγκες του τομέα. Δηλαδή οι προτάσεις, η πρόταση ε, περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες, αλλά αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσει ελέγχου θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν στους διάφορους τομείς. Και η συνθήκη της Λισαβόνας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα πιο ευέλικτο τρόπο νομοθεσίας, νομοθέτησης. η Κομισιόν επουδενή δεν έχει σκοπό να προετοιμάσει αυτές τις κατεξιδότητες πράξεις απομονωμένα. Θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει συνένεση σε όλες τις προτάσεις και θα γίνει διαβούλευση. Τώρα, να απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις για τα διδάγματα τα οποία έχει βγάλει η Κομισιόν από το σκάνδαλο για το ε, κρέας αλόγων. Κάναμε την αξιολόγησή μας και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και καινούρια κεφάλαια. Για παράδειγμα, Και εδώ απαντώ στο κατά πόσον η επίσημη έλεγχη είναι διαφορετική από τους ε, ελέγχους για τις απάτες. Υπάρχει το άρθρο 8, στο οποίο προστίθεται μία απέτηση από τα κράτη-μέλη. Στο πολιετές πρόγραμμα ελέγχων θα πρέπει να περιλαμβάνουν πλέον και ένα κεφάλαιο για τους ελέγχους ε, περί των ε, σκοπίμων ε, παραβιάσεων. Ξέρω ότι τα κράτη-μέλη επισκέφτονται τις, ε, μάλλον κάνουν ελέγχους ε, για να διαπιστωθεί το κατά πόσον γίνονται σεβαστοί γενικοί κανόνες, αλλά αυτή η έλεγχη δεν είναι αρκετή για να καταπολεμηθεί η απάτη. Γι' αυτό το λόγο λέμε στα κρατη ότι θα πρέπει να γίνονται ειδικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό της απάτης και να δίνεται και ειδική επιμόρφωση στους ελεγκτές. Δηλαδή δεν θα πρέπει να ελέγχονται μόνο τα εγγραφά, ε, για το κατά ναι, να γίνει τη διασταύρωση μεταξύ των ζώων που μπαίνουν και των ζώων που βγαίνουν. Δεν αρκεί αυτό. Επίσης έχουμε προσθέσει και μια ακόμα υποχρέωση στις, ε, στο κεφάλαιο ε, των ποινών, των κυρώσεων. Αυτό αφορά το ύψος των κυρώσεων για περιπτώσει απάτης. Θα πρέπει αυτό να είναι τουλάχιστον τόσο υψηλό όσο το κέρδος το οποίο θα προέκυπτε από την ίδια την απάτη. Γι' αυτό το λόγο είναι αποτρεπτικό. Μια άλλη αλλαγή προέκυψε μετά το σκάνδαλο ε, ήταν ε, να γίνουν υποχρεωτικά τα συντονισμένα σχέδια ελέγχου. Ε, είχαμε ζητήσει ε, τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τέτοιου είδους ε, σχέδια για τον εντοπισμό ε, κρέας αλόγου που δεν έφερε την κατάλληλη σήμανση. Αυτά τώρα τα σχέδια γίνονται υποχρεωτικά. Όταν γίνουν λοιπόν αυτά τα συντονισμένα σχέδια, θα είναι υποχρεωτικά, δηλαδή όταν γίνουν δεκτά θα, γίνουν, θα είναι υποχρεωτικά. Επίσης, έχουμε ε, διευκολύνει την διοικητική συνεργασία. Πολλά έχουν να γίνουν, πολλά είναι να γίνουν ακόμα ε, σε ό,τι αφορά την συνεργασία για την ε, καταπολέμηση απάτης διασυνοριακά. Η διασυνοριακή έλεγχη μπορεί να, γίνει, να είναι αποτελεσματική μόνο όταν οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται, μιλούν μεταξύ τους, τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα τα γεγονότα. Για παράδειγμα, ανταλλαγή πληροφοριών και συνδρομή έτσι ώστε να γίνει κατοδοτή η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας. Και πάλι επιστρέφω τώρα στη, στο θέμα των κατεξιότητας πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων. Αυτές οι εξουσίες ενδεχομένως θα μπορέσουν να βοηθήσουν και στην αντιμετώπιση ε, σκανδάλων τέτοιου τύπου γιατί θα μας έδιναν τη δυνατότητα η ε, οι στο μέλλον για συγκεκριμένους τομείς της ε, διατροφικής αλυσίδας να γίνουν πιο ομοιόμορφοι και θα έδιναν τη, τη δυνατότητα ε, στα, στην Κομισιό να πει στα τι γίνεται με το μη χνηλατημένο κρέας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια, κατακαιρματισμένη, μια προσέγγιση και ενδεχομένω χρειάζεται να την ε, κάνουμε πιο ομοιόμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mrs. Um, Ευχαριστώ κυρία Γκαρό. Ζητούν ε, κάποιοι το λόγο για να κάνουν και άλλες ερωτήσεις. Να, να δώσω όμως το λόγο στον εισηγητή κύριο Πυρίλο, γιατί είπε ότι πρέπει να προλάβει κάποια στιγμή μια πτήση. Έχετε το λόγο κύριε Πυρίλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ άπαντες ε, για όλα τα σχόλια. Εμπλούτησαν ε, αυτές οι προτάσεις στη δική μου έκθεση. Συμφωνώ με ορισμένες προτάσεις. Κάποιες άλλες θεωρώ ότι θα πρέπει να τις εμβαθύνουμε περισσότερο. Με απασχολεί λίγο η πρόταση για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό. Θα πρέπει να το εμβαθύνουμε. Αναμφίβολα, αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να μας ξεφύγει. Μπορεί να μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε πιο ακριβείς ελέγχους των προϊόντων διατροφής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και την Κομισιόν και πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε και να συνεργαστούμε στο μέγιστο και με τα κράτη-μέλη. Αυτό θα μας βοηθήσει να βγούμε από κάποιες περίπλοκες καταστάσεις ε, όπως τις συζητήσαμε σήμερα το πρωί, τις υποδείξαμε σήμερα το πρωί, αλλά πιστεύω ότι με τις τροπολογίες που θα υποβάλουμε στις επόμενες συναντήσεις ε, σίγουρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα ώστε ο κανονισμός αυτός να μπορεί να εφαρμοστεί έγκαιρα και σωστά από τα κράτη-μέλη ώστε να αποφευχθούν οι διαφορετικές εφαρμογές και οι διαστρεβλώσεις μεταξύ κρατών μελών. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πυρίλο για τις τελευταίες παρατηρήσεις. Εδώ κλείνουμε το σημείο 4. Προθεσμοί για τροπολογίας είναι 12 Δεκεμβρίου, 12 η ώρα και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 30 Ιανουαρίου του 2014. Αυτό μας φέρνει στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση του Μπαρτστάς για τις μεταφορές αποβλήτων. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Σεγητή, τον Μπαρτστάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να προτείνω κάτι άλλο. Συμφώνησα με την Κομισιόν να μιλήσουν αυτοί πρώτα, να μας κάνουν μια εισαγωγή και μετά να λάβω εγώ το λόγο. Θα προτιμούσα λοιπόν να δώσουμε το λόγο στη Κομισιόν πρώτα. Thank you, uh, Chair. Um, I will then give a... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να κάνω μια σύντομη εισαγωγή για αυτή την πρόταση σε τρία μέρη. Πρώτα απ' όλα ποιο είναι το πρόβλημα, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόταση. Δεύτερον για ποιο λόγο έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και τρίτον τι προσπαθεί να κάνει η πρόταση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Τώρα όσον αφορά το ποιο είναι το πρόβλημα. Μιλάμε για τις παράνομες μεταφορές αποβλήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς άλλα μέρη του κόσμου. Κυρίως στην Αφρική και την Ασία. Έχουμε αναφορές που μας λένε ότι πρόκειται για σημαντικό ποσότητες, ε, σημαντικό ποσοστό των μεταφορών αυτών είναι παράνομος. Παράνομος σημαίνει πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα τίθεται το ζήτημα διάκρισης μεταξύ εμπορευμάτων και αποβλήτων. Δεν είναι πάντα σαφές κατά πόσο μιλάμε για απόβλητα ή για αγαθά ή εμπορεύματα. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός αποστέλλεται σε τρίτες χώρες για επαναχρησιμοποίηση, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για απόβλητα και δεν μπορούν να, που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Υπάρχει λοιπόν το ζήτημα αυτής της διάκρισης. Δεύτερον, εάν ένα πλοίο μεταφέρει τα απόβλητα για ανάκτηση σε κάποια τρίτη χώρα, για ανακύκλωση. Δεν ξέρουμε αν όντως καταλήγει σε εγκαταστάσεις ανακύκλωση σε τρίτη χώρα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ζήτημα διάκριση μεταξύ ανάκτηση ανακύκλωση ή διάθεσης. Απόρριψη, δηλαδή. Πρώτος στόχο λοιπόν της πρόταση αυτής ε, είναι προφανώς ε, να διασφαλίσουμε το περιβάλλον και τη δημοσία υγεία στις τρίτες χώρες. Παρέχει επίση ένα οικονομικό όφελος διότι όταν αποστέλλονται παράνομα απόβλητα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωση, πρέπει να επαναπατριστούν και αυτό κοστίζει πολύ. Επίσης και το κόστος καθαρισμού και των ζημιών προς τρίτες χώρες είναι πολύ ψηλό. Συνεπώς οι παράνομες αυτές δραστηριότητες μπορεί να έχουν πολύ ψηλό κόστος. Επίσης ε, βοηθά στη διατήρηση των πόρων εντός της Ευρώπης ε, η αποφυγή της παράνομης μεταφοράς αποβλήτων σημαίνει ότι η ανακύκλωση και η επανάχρηση μπορούν να γίνουν στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο έχουμε αυτό το πρόβλημα. Κυρίως διότι οι δυνατότητες επιθεώρησης εμπορευμάτων, αποβλήτων, μεταφορών γενικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλές περιπτώσεις ε, παρουσιάζει ελλείμματα. Κάποια κράτη-μέλη έχουν πολύ καλά συστήματα επιθεώρησης Αλλά όπως τεκμηριώνεται στις μελέτες που κάναμε σε πολλά κράτη-μέλη δεν υπάρχει προγραμματισμός των επιθεωρώσεων. Οι πόροι που χρησιμοποιούνται για τις επιθεωρήσεις είναι ελάχιστοι. Και έτσι λοιπόν πολλά πλοία φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από λιμάνια κρατών μελών με πολύ χαμηλό έλεγχο Υπάρχει αυτό το φαινόμενο του port hopping, της αποφυγής λιμένων, ε, δηλαδή φεύγουν τα πλοία αυτά από τα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρήσει είναι ελάχιστες. Επίσης έχουμε πρόβλημα διότι, έχουμε το πρόβλημα αυτό διότι το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις αποστολές εμπορευμάτων και αποβλήτων δεν το ρυθμίζει με ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Υπάρχει το άρθρο 50 που μιλάει για επιθεωρήσεις αλλά αναφέρεται σε αυτές γενικά δεν λέει πραγματικά στα κράτη-μέλη τι πρέπει να κάνουν όσον αφορά τις επιθεωρήσεις και τον προγραμματισμό τους. Εμείς ε, πραγματοποιήσαμε μια μεγάλη διαβούλευση ενδιαφορμένων όπου διαπιστώσαμε μεγάλη υποστήριξη από τη βιομηχανία της ΜΚΟ και λοιπούς ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να ενισχύσουμε τις απαιτήσει ε, προγραμματισμού των επιθεωρήσεων. Περνώ τώρα στο τρίτο κομμάτι, τι προτείνουμε να γίνει σε αυτή την πρόταση. Προτείνουμε τροποποίηση ή συμπλήρωση του υπάρχοντος άρθρου 50 στο κανονισμό περί αποστολών εμπορευμάτων. Το άρθρο 50 αυτό μιλάει για επιθεωρήσεις μόνο γενικά. Η πρόταση απαιτεί από τα κράτη-μέλη να καθιερώσουν σχέδια επιθεωρήσεων για εμπορεύματα, γενικώ αποστολές, μεταφορές εμπορευμάτων ορίζει μια σειρά ελάχιστον υποχρεωτικών ε, στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνουν τα σχέδια αυτά, σαφείς στρατηγικούς στόχους, χρήση αξιολόγησης επικινδυνότητας, ώστε να εντοπίζονται οι κύριοι σοδοί ε, παρανομής μεταφοράς, να οριστούν προτεραιότητες πληροφορίες σε σχέση με τη φύση και τη συχνότητα των επιθεωρήσεων αποβλήτων ή αποστολών, τη δέσμευση επαρκών πόρων, την ενημέρωση σε σχέση με τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων λιμενικών αρχών και την πρόβλεψη απαραίτητης κατάρτισης των επιθεωρητών. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο της πρότασης. Το δεύτερο στοιχείο της πρότασης είναι ότι πιστεύουμε πως είναι πολύ σημαντικό τα σχέδια αυτά επιθεωρήσεων να είναι δημόσια. Να υπάρχει λοιπόν υποχρέωση δημοσίευσης των σχεδίων αυτών, ώστε το κοινό να γνωρίζει, ο κόσμος να γνωρίζει ότι οι επιθεωρήσεις λαμβάνονται σοβαρά και ότι τα κράτη-μέλη πραγματικά κάνουν κάτι αυτό για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τρίτον, το τρίτο στοιχείο της πρότασης είναι ότι σε περίπτωση υποψίας παράνομων αποστολών είτε γιατί υπάρχει υποψία ότι η αποστολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάλλον απόβλητα και όχι εμπορεύματα είτε διότι υπάρχει υποψία ότι κάποιο εμπόρευμα ή κάποια απόβλητα που φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα καταλήξουν σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αλλά θα διατεθούν σε χώρους απορριμμάτων οι αρχές πρέπει να αποδείξουν ότι το φορτίο που φεύγει είναι όντως απόβλητα και μπορούν να ζητήσουν αποδείξεις, αποδεικτικά στοιχεία για τον προορισμό των αποβλήτων ώστε να είναι βέβαιες ότι πράγματι καταλήγουν σε εγκαταστάσεις ανάκτησης και ότι δεν αποτίθενται κάπου παράνομα. Το τέταρτο στοιχείο είναι η τυπική ευθυγράμμιση επιτροπολογίας όπου έχουμε τη μεθοδο εξέταση. Προτείνουμε να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις αυτές της επιτροπολογίας με κατεξοδότηση πράξης. Αυτή είναι συνοπτικά η πρότασή μας. Ουσιαστικά θέλουμε τροπολογία του κανονισμού αποστολής αποβλήτων με τροπολογία του άρθρου 50. Το άρθρο αυτό υπάρχει, απλά θέλουμε να γίνει πιο συγκεκριμένο όσον αφορά τις απαιτήσει ε, που θα έχουν τα κράτη-μέλη για την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λάγκεντορφ, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δίνω το λόγο πάλι στον Μπαρτσάς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ε, έλαβα, ε, στην έκθεσή μου μάλλον έλαβα υπόψη ε, την ε, έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου των Κάτω Χωρών για το πώς εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία στην Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Σλοβενία, Νορβηγία και κάτω χώρε. Είναι ένα έγγραφο, μια έκθεση που κάνει πολλές παρατηρήσεις για το ε, πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία, περιλαμβάνει πολλές συστάσεις οι ε, θα ήθελα να συμπεριλάβω. Επίσης ε, επισκέφθηκα με τον ε, εισηγητή της Επιτροπής των Περιφερειών, τον Λιμένα της Ανβέρσας, που ήρθε σε επαφή με τελωνιακούς και με αστυνομικούς. Μίλησα με τους ελεγκτές της επιχείρησης διαχείρισης αποβλήτων, του, Βελγίου και των κατοχωρών. Ε, επίσης ήρθα σε επαφή ε, είδα μάλλον ένα μικρό σποτ το οποίο παρουσιάζει το έργο των ε, επιθεωρητών ελεγκτών. Οι επιθεωρητές ε, είχαν μάλιστα εντοπίσει δύο υποψίες για ένα φορτίο από την Αφρική και ένα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν ανοίξαμε τα κοντέινερς, κοιτάξτε τι ανακάλυψαν. Je Όπως βλέπετε, αυτό είναι το φορτίο που ερχόταν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπήρχαν μικρά φορτηγάκια που ήταν γεμάτα ε, με απόβλητα από αυτοκίνητα, μεταχισμένα αυτοκίνητα, ε, παλιού, παλιά πεταμένα ψυγεία, παλιές καρέκλες. Ο εισηγητής Επιτροπής των Περιφερειών ήταν ε, Βρετανός και ζήτησε συγγνώμη για το γεγονό ότι τα φορτίο προερχόταν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω πως ε, άξιζε τον κόπο να σας προβάλλουμε αυτό το σποτάκι για να καταλάβετε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ε, μίλησα με τους ελεγκτές και χαίρονται πολύ για την πρόταση της Κομισιόν. Πιστεύουν όμως ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να βελτιωθούν. Εγώ εστίασα σε πέντε πράγματα. Πρώτον, πρέπει να βελτιωθεί η βάση γνώσεων σχετικά με τις παράνομες μεταφορές. Δεύτερον, ε, περιλαμβάνοντας τα σχέδια επιθεωρήσεων ένα ελάχιστο αριθμό υλικών, να, να περιλάμβουμε στα σχέδια επιθεωρήσεων ένα ελάχιστο αριθμό υλικών ελέγχων. Τρίτον, ε, η μόνιμη διάθεση στο κοινό των σχεδίων επιθεωρήσεων και των αποτελεσμάτων. Τέταρτον, εκχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων στις σχετικές αρχές. Και πέμπτον, βελτίωση συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης προτείνω και καινούριου ορισμού στο κείμενο, για παράδειγμα την επαναχρησιμοποίηση, βασίζομαι στην οδηγία 2008-98, καθώς επίσης και τον ορισμό των ελέγχων. Σε ό,τι αφορά το πρώτο από αυτά τα πέντε σημεία, δηλαδή η βάση γνώση σχετικά με τις παραδιαταφορές, όλοι όσοι ε, μου μίλησαν καθώς επίσης και η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, λένε πως χρειάζεται ένα εναρμονισμένο πρωτόκολλο για την καταγραφή των ε, δεδομένων αυτών, των δεδομένων των ελέγχων. Χρειάζεται επίσης ε, ένας ε, πίνακας μετατροπής μεταξύ τελωνιακών κωδικών και κωδικών των αποβλήτων. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να γίνει σύγκριση. Χρειάζονται επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποινικοποίηση των παρεμβάσεων ε, και ασφαλώς χρειάζεται και εναρμόνιση σε αυτό το τομέα. Γνωρίζουμε ότι όταν οι ποινέ διαφέρουν, οι διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ε, γίνεται ε, όλες οι παράνομες συναλλαγές ε, περνούν από συγκεκριμένα λιμάνια. Δεύτερον, ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να περιλαμβάνουν ένα ελάχιστο αριθμό φυσικών ελέγχων των εγκαταστάσεων και των μεταφρών αποβλήτων σύμφωνα με τη στρατηγική και τους στόχους, καθώς και μια αξιολόγηση του κινδύνου που, έχει, που, διενεργείται προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο επιθεωρήσεων. Τρίτον, είναι σημαντικά τα σχέδια επιθεωρήσεων να είναι μονίμως στη διάθεση του κοινού. να πω ότι ορισμένοι θεωρούν πως ε, ότι δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά ε, ελεγκτικοί Γι' αυτό εγώ μιλώ για επιχειρησιακά σχέδια τα οποία δεν θα ε, δημοσιεύονται, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα στοιχεία τα οποία ε, είναι δυνατόν να τα δημοσιεύουμε, να έχει προσβαστεί το κοινό, χωρίς να δίνουμε στοιχεία στους ε, παρανομούντες έτσι ώστε να ξεφύγουν από τους ελέγχους. Ο εκπρόσωπος Κομισιόν το είπε ότι τέτοιου είδους πληροφορίες, δημόσιες πληροφορίες ε, έχουν θετικό αντίκτυπο. Τέταρτον, το σημείο στο οποίο ε, εστίασα, εκχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων στις σχετικές αρχές. Αυτή τη στιγμή ε, θεωρούμε ότι ορισμένες υπηρεσίες ή μάλλον ορισμένες νομοθεσίες κρατών μελών, για παράδειγμα του Βελγίου, προβλέπουν ότι ε, δεν χρειάζεται να υπάρχει υποψία για να γίνει έλεγχος. Όμως σε άλλες νομοθεσίες δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται μόνο όταν υπάρχουν υποψίες. Ε, λοιπόν, εγώ προτείνω πράγματι να διαγραφεί, να καταργηθεί η υποχρέωση ύπαρξης υποψίας. Μετά, πέμπτο σημείο, συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. συνεργασία μεταξύ κρατών μέλων είναι απολύτω απαραίτητη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίε για τι μεταφορέ αποβλήτων. Αυτή τη στιγμή γίνονται, μεταφορές, γίνονται ανταλλαγέ πληροφοριών, αλλά μόνο σε επίπεδο ad hoc, σε επίπεδο προσωπικών γνωριμιών. Δεν είναι κάτι υποχρεωτικό και δεν υπάρχει και ένα ενιαίο σύστημα. Θα πρέπει οι ανταλλαγές να γίνουν με ε, στο κατάλληλο πλαίσιο, να είναι υποχρεωτικές, τακτικές και διαρθρωμένες. Νομίζω ότι η Κομισιόν θα μπορούσε να πάρει μια πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτές είναι οι βασικές μου προτάσεις. Σε ό,τι αφορά την επιτροπολογία, Προτείνω την ευθυγράμμιση όλων των υφιστάμενων διατάξεων ε, επιτροπολογίας με το άρθρο 290 προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή ε, αντί να καλυφθούν επιμέρους σημεία μέσω της ε, πρότασης Omnibus. Προτείνω οι τροπολογίες να κατα... υποβληθούν μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Θα έρθω σε επαφή με τους κοιόδης ηγητές στο Στρασβούργο. Και το Δεκέμβριο, ενδεχομένω και τον Ιανουάριο, έτσι ώστε να ψηφιστεί πρώτα τη βδομάδα τη 23 η Ιανουαρίου. Είμαι σε επαφή και με το Συμβούλιο, με την ε, σημερινή Προεδρία και θα έρθω σε επαφή και με την επόμενη Προεδρία έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε να έχει κλείσει το θέμα πριν λήξει η θητεία μας. Με ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο Καρλ Χάινς Φλόρενς. Ευχαριστώ νομίζω έκανες πολύ καλή πρόταση και η Κομισιόν έκανε το καλύτερο δυνατό και εγώ δεν θα αντιταχθώ σε όλα αυτά αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι ε, όλα αυτά είναι και λίγο ε, λυπηρά με τα κράτη-μέλη που δεν θέλουν να τους προδιαγράφουμε τι να κάνουν και τι να μην κάνουν. Και βλέπουμε εδώ στις εξαγωγές αποβλήτων ότι πολλές χώρες και οι δικοί μου δεν κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους. Η αντίδρασή μας πια είναι περισσότερη γραφειοκρατία. Βέβαια ομολογώ ότι και εγώ καλύτερη λύση δεν έχω, αλλά είναι ντροπή. Από τη μία πλευρά μας επιτίθενται ότι έχουμε υπερβολικά πολλές διατάξεις και από την άλλη τα κράτη-μέλη δεν μπορούν καν πρώτες ύλες που είναι ε, κληροδότημα των παιδιών μας να τις διαχειρίζονται σωστά. Πρέπει να μιλάμε με περισσότερα ονόματα, πιστεύω, γιατί εδώ είμαστε σαν όμιλος που δεν αναφέρει ονόματα νομίζω ότι ε, οι πρεσβευτές των χωρών που επιδεικνύουν αμέλεια θα έπρεπε να ε, εγκαλεστούν. Και αυτό δεν γίνεται. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάνουμε σχέδια, καταλόγους ελέγχων, γι' αυτό χρειάζεται βέβαια να υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό, διαθέσιμη πόροι και γιατί όλα αυτά, γιατί τα κράτη-μέλη δεν ανταποκρίνονται στο έργο που τους έχει ανατεθεί. Δεν ε, ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που έχουν. Και ε, μου κάνει εντύπωση η υπομονή που, με την οποία αντιμετωπίζομαι την αμέλεια πολλών ε, υπεύθυνων στα κράτη-μέλη και πάμε να τα καλύψουμε. Αυτό είναι σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ούτω ώστε επιτέλους σε κοινοτικό επίπεδο μάλλον σε επίπεδο κρατών μελών αποφασίζεται αυτό που αποφασίσαμε σε ενωσιακό επίπεδο. Ε, φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη μας ε, δεν έχουν την ε, υπευθυνότητα που απαιτείται για κάτι τέτοιο. Η συνάδελφος Λούμπετσεβα. Ευχαριστώ. Αυτή η έκθεση αφορά με το, αφορά τον κανονισμό για τις εξαγωγές αποβλήτων και είναι ένα καλό παράδειγμα σχετικά με το τι κάνει στον τομέα του περιβάλλοντος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές ότι υπήρξαν πολλές παρατυπίες εις ό,τι αφορά τις μεταφορές αποβλήτων. Και ε, το ποσοστό είναι 25 με 50% των μεταφορών αποβλήτων που δεν ανταποκρίνεται στις ε, διατάξεις. Δύο σημαντικά πράγματα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εδώ. Τον οικονομικό παράγοντα τι και τους κοινωνικούς πόρους και όποτε υπάρχουν παρατυπίες δεν κερδίζει κανείς. Παράλληλα είναι σημαντικό να τονίσουμε την επίπτωση όλων αυτών στη δημόσια υγεία. Είναι λοιπόν σαφέστατο ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι σε θέση να λύσει το πρόβλημα των παρατυπιών στις μεταφορές αποβλήτων σωστά. Υπάρχουν δε πολλές διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Γι' αυτό χρειάζεται η τροποποίηση αυτού του κανονισμού και θα πρέπει να προσθέσουμε κι άλλες απαιτήσει σχετικά με την μεταφορά αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Και εις ό,τι αφορά τις τροπολογίες και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε τον εισηγήτη για την έκθεση. Καταρχήν που συμφωνώ. Πρώτον, είναι σαφέστερες ε, οι διαδικασίες σχετικά με τους ελέγχους. Επίσης, ο προορισμός των αποβλήτων παρακολουθείται πολύ προσεκτικότερα. Οι διαδικασίες για την κοινοποίηση επίσης απαιτούνται και όποτε διαπιστώνονται παρατυπίες ενημερώνεται και η κοινή γνώμη. Οπότε η πρόταση είναι πολύ καλή. Επίσης η Κομισιόν μπορεί να θεσπίσει κατεξουσιοδότηση πράξης σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων. Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μία ισορροπία ε, μεταξύ των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των κατεξουσιοδότηση πράξεων που θεσπίζει η Επιτροπή. Νομίζω ότι η έκθεση είναι πολύ ισορροπημένη και συμβάλλει στην ποιο... Ε, εφαρμογή των ποιοτικών προτάσεων της Κομισιόν και διευκρινίζει ορισμένα θέματα. Είναι σαφείς οι στόχοι που καταγράφονται και αφορούν στην περιβαλλοντική προστασία, και την ε, κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ε, οικείων θεσμικών οργάνων και θεσμών. Γι' αυτό γενικά συμφωνούμε ότι πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός και θα καταθέσουμε και ε, τροπολογίες για να παρουσιάσουμε τις προτιμήσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Thank um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε την τηλεοπτική σειρά ε, The Sopranos για την οικογένεια της μαφίας και ε, ρώτησαν τον Τόνι Σοπράνο τι κάνει, τι δουλειά κάνει και έλεγε ότι είναι σύμβουλος διαχείρισης αποβλήτων. Και παρά το γεγονό ότι η βιομηχανία αποβλήτων γίνεται όλο και πιο επαγγελματική, αν δείτε τα νούμερα στα έγγραφα της Κομισιόν, περίπου το 25% των ε, αποστολών ε, αποβλήτων παραμένει παράνομη. Παρότι έχει αποβίωσει πριν από λίγου μήνε ο ηθοποιό που έπαιξε τον Τόνι Σοπράνο, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί Τόνι Σοπράνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να καταπολεμήσουμε για πολλού λόγου αλλά να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Μπάρτ Στάς για την εξαιρετική του έκθεση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εκπληκτικό του έργο. Το τομέας αυτός ε, μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Πρέπει να καταλήξουμε γρήγορα σε κάποια συμπεράσματα να βελτιώσουμε την νομοθεσία το ταχύτερο δυνατόν. Υποστηρίζω λοιπόν τον Μπαρτιστάς ε, στο φιλόδοξο χρόνο του και στις προσπάθειες του να προσπαθεί να επιτύχει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση πριν από τις ευρωεκλογέ του χρόνου. Για μένα το σημαντικότερο, πέραν του γεγονότος ότι μιλάμε για παράνομες δραστηριότητες, είναι και η απόδοση των πόρων, η αποδοτική χρήση των πόρων. Παρατηρούμε αποστολή πολύ σημαντικών πόρων εκτός Ευρώπης, παράνομα πόρους τους οποίους χρειαζόμαστε απελπισμένα. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να τους ανακτήσουμε. Υποστηρίζω επίσης τον Παρθάς απολύτως ε, στη σύνδεση που κάνει μεταξύ αυτής της οδηγίας αποστολής ε, αποβλήτων και της οδηγίας ε, των ηλεκτρονικών συσκευών Είναι σημαντικό επίσης να επεκτείνουμε τους τομείς ε, όπου υπάρχει δυνατότητα επιθεώρησης ε, από τους επιθεωρητές, όχι μόνο στις αποστολές, αλλά και στις ε, εγκαταστάσεις συλλογής, περισυλλογής και αποθήκευσης. Σύμφωνα με τις μελέτες, το 80% των επιχειρήσεων δεν συμμορφώνονταν με τους κανόνες, όπως διαπιστώθηκε από επιθεωρήσεις στους χώρους τους. Μπορούν λοιπόν να γίνουν πολλά και εκεί. Τώρα, όσον αφορά τη δημοσίευση των σχεδίων επιθεώρηση. συμφωνώ με τον Καρλ Χάιντς Φλόρεντς ε, ε, από τους σοσιαλιστές. Ε, πρέπει να προσέχουμε τη γραφειοκρατία. Μίλησα με κάποιους επιθεωρητές και αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα επηρεαστούν από την επιπλέον γραφειοκρατία. Αυτοί ζητούν δημοσίευση των σχεδίων επιθεώρησης διότι τους είναι απαραίτητα στο έργο τους, στην καταπολέμηση των παράνομων αποστολών. Πιστεύω λοιπόν ότι το θέμα εδώ δεν είναι η γραφειοκρατία. Το θέμα είναι να βρούμε έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο διεξαγωγής των επιθεωρήσεων. Έχω να πω πολλά, αλλά θα επαναλάμβανα τα όσα είπαν ο Μπαρτιστάς, η Κομισιόν και όλοι οι άλλοι ομιλητέ ήδη. Δυο τελικά σχόλια εκ μέρους μου κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, η θέση των πληροφοριδοτών, των whistleblowers. Η αγορά αυτή είναι πολύ περίεργη. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν ε, κατά πόσο οι πληροφοριοδότες ε, εντός της βιομηχανίας προστατεύονται επαρκώς αυτή τη στιγμή κατά πόσο θα πρέπει να προβλέψουμε κάποιες διασφαλίσεις για αυτούς. Και η τελευταία παρατήρηση και οι πληροφορίε μου έρχονται από επιθεωρητέ. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλέ συναλλαγέ σε μετρητά στην αγορά αυτή. Σε κάποια με λίγα απαγορεύονται. Στι κάτω χώρε, στη δική μου χώρα δεν απαγορεύονται. Υπάρχουν πολλέ συναλλαγέ λοιπόν σε μετρητά. Και αυτό δυσχεραίνει το έργο των επιθεωρητών. Επίσης ε, δίνει και μια σκιώδη εικόνα κάπως της ε, αγοράς αυτής. Ε, είναι εύκολο να καλύψει κανείς παράνομες μεταφορές. Αυτή είναι λοιπόν μια άλλη μου ερώτηση προς την Κομισιόν. Πιστεύει η Κομισιόν ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μήπως θα έπρεπε να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο για να πείσουμε τα κράτη-μέλη να φροντίσουν να διακοπούν αυτές οι συναλλαγές μετρητά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Ιάννα Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Στάση και την ε, Κομισιόν εκ μέρους της ομάδας μου. Η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει. Και πιστεύουμε ότι η Κομισιόν βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Όμως υπάρχουν και κάποιες αδυναμίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και επιβολή του νόμου και τις διαφορές στην εφαρμογή του νόμου μεταξύ χωρών. Η έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις ε, θα πρέπει να είναι ευνηδιαστικοί, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί. Τα απόβλητα πλέον δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεφορτωθούμε είναι πόροι οι οποίοι μπορούν να ε, τύχουν επανεπεξεργασία στην Κομισιόν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να εξάγουμε τα απόβλητά μας και ιδιαίτερως δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να τα εξάγουμε παράνομα. Η ε, εκμετάλλευση των αποβλήτων μπορεί να γίνει προς οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει οι παράνομες εξαγωγές αλλά και οι γενικότερα εξαγωγές να ε, καταργηθούν. Επίσης θα πρέπει να τηρούμε πάντοτε την αρχή της επικουρικότητας. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να παραχωρήσουμε στην Κομισιόν περισσότερες εξουσίες από αυτές που χρειάζεται. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή για αυτό το πολύ καλό σχέδιο έκθεσης. Περιμένω θα συνεργαστούμε επικοδομητικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τέλος ο εισηγητής Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Γκαϊμπαντή ρώτησε κάποια πράγματα στην Κομισιόν. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να μην ξεχάσουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις της Κομισιόν. Θα ήταν χρήσιμο. Βλέπω ότι υπάρχει ευρεία υποστηρίξη για την πρότασή μου. Πολύ ευχάριστο αυτό. Τώρα για τα είπε ο κύριος Φλόρεντς, αυτή η ιδέα της κατονομασίας του naming and shaming. Σίγουρα δεν κατανομάζεται ονόματα, αλλά νομίζω θα πρέπει να κάνουμε μια συνάντηση με τους Κιώδες ίσως ε, για να καταρτήσουμε έναν κατάλογο των ε, κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται στο μεγαλύτερο βαθμό. Θα ήταν καλή ιδέα αυτή. Και μετά θα μπορούσαμε να συντάξουμε μια επιστολή προς τις μόνιμες αντιπροσωπίες των κρατών μελών αυτών, ώστε να τους ζητήσουμε εξηγήσει θα μπορούσαμε να το πράξουμε αυτό εντός του νομοθετικού πλαισίου ως μια ε, ειδοποίηση προς τα κράτη-μέλη. Νομίζω καλή θα ήταν η ιδέα αυτή και ευχαριστώ τον κύριο Φλόρεντς που έθεσε το θέμα αυτό. Όσον αφορά τα υπόλοιπα σχόλια, εγώ προτείνω το εξή Να εστιαστούμε στην βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ αρχών επιθεωρήσεων δεν νομίζω ότι τίθε θέμα γραφειοκρατία εδώ, το είπε και ο κύριο Γκεμπράντη. Αυτό ακούω και από τι ίδιε τη υπηρεσία επιθεωρητών. Θέλουν καλύτερη και περισσότερη συνεργασία, περισσότερη δημοσιοποίηση των πληροφοριών και κοινοποίηση των πληροφοριών γιατί του επιτρέπει να διεξάγουν το έργο του πιο αποτελεσματικά. Οι ίδιοι το ζητούν. Του βοηθούν οι στενότερε επαφέ με του συναδέλφου του. Θα κλείσω εδώ. σω θα μπορούσε η Κομισιόν όμω να απαντήσει τι ερωτήσει που έγιναν προς αυτήν. Ευχαριστούμε Κομισιόν. Πριν προσπαθήσω να πω κάτι για αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα και να δώσω απαντήσεις, να πω δύο λόγια για την ίδια την έκθεση, αν δεν έχετε αντίρρηση. Είμαστε φυσικά ικανοποιημένοι που η έκθεση, το σχέδιο έκθεσης υποστηρίζει τα βασικά στοιχεία της πρότασής μας. Πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό ότι χωρίς να μπαίνουμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες για τις επιθεωρήσεις αυτές, ε, έχουμε κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις και προσπαθούμε να επιτύχουμε μια ισορροπία Ωστόσο, θεωρούμε ότι αν πρόκειται να υπάρξει απέτηση σχεδίων επιθεωρήσεων για τα κράτη-μέλη, αυτή η απέτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από μια σειρά υποχρεωτικών ε, στοιχείων, υποχρεώσεων, οι οποίες υποχρεώσεις δεν μπορούν να είναι επιλογές, δεν μπορούν να είναι προαιρετικές. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί στην έκθεση επίσης. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την υποστήριξη για την ε, κοινοποίηση των σχεδίων. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τους λόγους που εξέθεσε ο εισηγητής. Όσον αφορά την κατονομασία των name and shame ε, στην εκτίμηση επιπτώσεων ε, που συνοδεύει αυτή την πρόταση θα δείτε και τις καλές πρακτικές που έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βέλιο, στις κατοχώρες μέσω διαφόρων επιθεωρήσεων και σχεδίων επιθεωρήσεων και μπορείτε να εξέχετε τα δικά σας συμπεράσματα από τις βέλτιστες πρακτικές αυτές σε σχέση με τις λιγότερο καλές πρακτικές σε άλλα κράτη-μέλη. Καλό θα ήταν λοιπόν να το μελετήσετε αυτό. Τώρα όσον αφορά τις ερωτήσεις που ακούσαμε, φοβάμαι ότι θα πρέπει να τις ε, μελετήσουμε οι πληροφοριοδότες, ε, οι whistleblowers. Νομίζω ότι δεν μπορούμε, πιστεύω, το θέμα αυτό να το αντιμετωπίσουμε σε αυτό τον κανονισμό για τη μεταφορά αποβλήτων. Το ίδιο και ισχύει και για τις συναλλαγές σε μετρητά. Θα τα μελετήσουμε και θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε μαζί σας τον τυχόν τρόπο αντιμετώπισης τους. Δεν είναι όμως κάτι εύκολο πιστεύω σε ένα τέτοιο νομοθέτημα για τη μεταφορά αποβλήτων να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και έτσι ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 3η Δεκεμβρίου ώρα 12. Στην 22-23 θα συζητήσουμε, τον Ιανουάριο θα συζητήσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για την έκθεση και ε, Μάρτιο-Απρίλιο 2014 θα συζητήσουμε την έκθεση στην Ολομέλεια. Προχωρούμε με το σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη. Ψάχνω την εισηγήτριά μας. Ωραία. Τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, στον ΕΟΦ. Η Λίντα Μακάβαν είναι η εισηγήτρια και θα λάβει πρώτη το λόγο. Λίντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη που βγήκα από την αίθουσα γιατί γίνονται πολλά ταυτόχρονα ε, στο νομοθετικό τομέα οπότε πρέπει να τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, ε, σήμερα θα μιλήσω για τις ε, τροπολογίες για τα τέλη φαρμακοεπαγρύπνησης. θα είναι πολύ γρήγορα γρήγορη συζήτηση, συμφώνησαν όλοι, έχουμε 100 τροπολογίες κατατεθειμένες στο Κοινοβούλιο, οπότε δεν είναι απλά τα πράγματα εδώ. Ξέρω ότι γίνονται πολλά και στο Συμβούλιο. Για να δούμε λοιπόν τις ε, τροπολογίες, θα ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις. Από συναδέλφους βέβαια οι περισσότεροι δεν είναι εδώ, αλλά θα τους στείλουμε σημείωμα για να διευκρινίσουν τι εννοούν. Και απογοητεύομαι που κάποια δεν είναι εδώ, που θα έπρεπε να είναι, γιατί υπέβαλαν τροπολογίες για θέματα κέρια στην νομοθεσία. Τέλος πάντων, αρχίζομαι με τα βότανα και τα ομοιοπαθητικά. Πολλές ε, τροπολογίες κατέθεσαν οι συνάδελφοι εδώ για να μειωθούν τα τέλη, να εξαιρεθούν συνολικά από την νομοθεσία και θέλω η Κομισιόν να διευκρινίσει για τους συναδέλφους το πεδίο εφαρμογής εδώ, διότι αυτό που περιλαμβάνεται στην ομοθέσια είναι μόνο εξουσιοδοτημένα ε, ε, βότανα, όχι τα καταχωρισμένα βότανα και ομοιοπαθητικά. Δηλαδή, ε, όταν επιλέξουν να κάνουν πλήρη κλινικό έλεγχο, ε, αυτά ε, ε, περιλαμβάνονται. Αυτά τα οποία είναι καταχωρημένα δεν είναι στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, οπότε αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Τώρα, για τα καταχωρημένα ομοιοπαθητικά, τα τέλη είναι τριών ειδών. Ε, είναι αυτά που είναι για τις, ε, το κεντρικό αποθετήριο ΠΕΑ, περιοδική επικαιροποιημένη, αυτά τα οποία είναι από τις εταιρείε ε, ομοιοπαθητικής και βοτανοθεραπευτικής, αυτά τα οποία είναι για τις μετεγκριτικές μελέτες και το καταποκοπήν τέλος. Κάποιοι λένε να μειωθεί το τέλος για τα βοτανοθεραπευτικά, ομοιοπαθητικά σε κάθε κατηγορία τέλους. Αλλά αν ένα βότανο θεραπευτικό ε, πρέπει να ε, υπόκειται σε περιοδική επικαιροποιημένη έκθεση ΠΑ. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να πληρώνουν ε, τέλος, γιατί έχουν δραστικές ουσίες, δεν είναι ουδέτερα προϊόντα και τα βοτάνο θεραπευτικά μπορεί να έχουν υψηλής δράσης, δραστική. Οπότε αν πρέπει να γίνει μια έκθεση επικαιροποιημένη, μια μελέτη, μου φαίνεται ότι και αυτοί πρέπει να πληρώνουν τέλος. 40-42 ε, τροπολογίες ε, εκεί ξέρουν τελείως από το τέλος ΠΕΑ ε, ή δίνουν μια έκπτωση 90%. Δεν ξέρω ποια είναι τα περιθώρια κέρδους όλων αυτών των εταιριών, δεν ξέρω πώς συγκρίνονται με τα κέρδη κάποιων μικρών φαρμακευτικών εταιριών, για παράδειγμα, αλλά θα ήθελα να σχολιάσει και εδώ η Κομισιόν. Τώρα, ένας αριθμός τροπολογιών επίσης προβλέπουν εξαιρέσεις για ε, εξουσιοδοτημένα ε, φάρμακα ομοιοπαθητικά από το ετήσιο τέλος ή τα εξαιρούν ολοσχερός. Θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν, πιστεύει ότι αυτό είναι δικαιολογημένο, πιστεύει ότι επειδή μάλλον τα ομοιοπαθητικά και βότανο-θεραπευτικά θέτουν λίγα θέματα φάρκα, φάρμακο επαγρύπνησης και δεν έχουν ε, πολλές παρενέργειες όπως αυτές που αναφέρονται εξαιρούνται, γιατί αυτό το ζητούν πολλοί συνάδελφοι που κατέθεσαν τροπολογίες για τα γενώσιμα τώρα. Τα γενώσιμα ε, ήδη ε, έχουν λιγότερες απαιτήσεις και η Κομισιόν λέει ότι 10 με 15% των δραστικών που χρήζουν ΠΕΑ ε, είναι γενώσιμα. Πρέπει, προβλέπει μείωση 20% από το ετήσιο τέλος για τα γενώσιμα η Κομισιόν. Εγώ το τροποποίησα αυτό ε, με βάση τις, ε, και τις τροπολογίες Ριβάζη και Ροτ Μπέρεντ, γιατί μειώσαμε το κάναμε ε, ε, 20% μείωση του καταποκοπήν, ε, γιατί αλλάξαμε τον υπολογισμό του ετήσιου τέλους. Λιγότερα μπαίνουν στη βάση δεδομένων ως γενώσιμα και κάναμε αλλαγή. Δεν παίρνουμε το μέγεθος της συσκευασία, αλλά το είδος της δραστικής. Τα γενώσιμα λοιπόν θα πρέπει λογικά να πληρώνουν λιγότερο, ε, με βάση τα προϊόντα, τον αριθμό των προϊόντων στη βάση δεδομένων. Επίσης είδαμε το πεδίο εφαρμογής του ετήσιου τέλους για να καλύψει ε, τις περιοδικές εκθέσεις. Όταν συμφωνήσαμε για τη φαρμακοεπαγρύπνηση, ο ΕΟΦ θα έπρεπε να κάνει παρακολούθηση πριν, πριν ε, προβεί στην ανάθεση αυτών των ε, υποχρεώσεων. Το ΕΟΦ λοιπόν θα παρακολουθούσε κοινέ ουσίες, πολύ κοινέ και πολλά, μου λένε ότι υπάρχουν πολλά γενώσιμα που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Ε, οπότε εδώ θα πρέπει να δούμε το θέμα της μείωσης του ετήσιου τέλους που αφορά κυρίως την παρακολούθηση των δεδομένων και το κεντρικό αποθετήριο ΠΑ και τη βάση δεδομένων αν έχουν πολλά προϊόντα στην αγορά. Κάποιοι συνάδελφοι εισάγουν νέα κατηγορία μείωση τελών για όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά εδώ και 10 χρόνια διότι οι καινοτόμε ε, βιομηχανίες λένε ότι δεν είναι δίκαιο να έχουν μείωση τα γενώσιμα ενώ τα δικά του να μην την χάνουν μείωση. Ε, και εδώ θα ήθελα το σχόλιο της Κομισιόν. Γιατί δεν το κάνατε. Είναι βιώσιμο, ε, είναι εφαρμοστέο, δηλαδή μπορεί να γίνει. Κάποιοι ζητούν μείωση για τις εταιρείε που αντιμετωπίζουν προβλήματα και αντιξοότητες. Σε αυτή την περίπτωση να έχουν έκπτωση και αυτοί. Εμένα δεν μου φαίνεται αυτό πολύ ε, ε, εφικτό, γιατί δεν είναι σαφές πόσο ο θα αποφασίσει ποιε θα είναι οι εταιρείε που έχουν να αντιμετωπίσουν αντικσότητες. Ε, κάποιοι μου λένε ότι πρέπει να μειωθεί το διοικητικό, ο διοικητικός φόρτος σε όλες τις νομοθετικές διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει δεν είμαι βέβαιη εδώ και να θυμόμαστε ότι θα πρέπει να δώσουμε λεφτά για να γίνει αυτή η δουλειά. Και αν όλοι έχουν έκπτωση και μειώσει στα τέλη, θα αυξηθεί το βασικό ποσό γιατί υπάρχουν κάποια χρήματα που πρέπει να είναι δεδομένα για να καλυφθεί το κόστος, για να έχουμε τη βάση δεδομένων, την παρακολούθηση και όλα αυτά που ζητάμε να γίνονται στην νομοθεσία και που θέλουμε να τα κάνει ο ΕΟΦ. Οπότε να μας εξηγήσει εδώ σαφώς η Κομισιόν παρακαλώ γιατί μειώσεις, ε, τι γνώμη έχει τις τροπολογίες, και τις αιτιολογήσεις τους. Οι συνάδελφοι δεν είναι εδώ βέβαια για να πούν οι ίδιοι πώς θα δικαιολογούν όλα αυτά. Ε, τώρα πλέον στα κράτη-μέλη. Ε, ε, κάποιοι έκαναν τροπολογίες που λένε πόσο πρέπει να πληρώνονται οι συνεισηγητές. Η Κομισιόν πρόβλεψε να αμείβονται και οι συνεισηγητές. Ε, και αν ναι, γιατί δεν λέτε στην πρόταση πόσα πρέπει να παίρνουν. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν βάλει αμοιβέ εισηγητών και συνεισηγητών τόσο ψηλέ που δεν μένει σχεδόν τίποτα για τον ΕΟΦ. Τι θα πάρει ο ΕΟΦ από τις αμοιβέ. Η Κομισιόν μπορεί να μας πει τι κάνει ο ΕΟΦ και ποιος είναι ο ρόλος του σε σχέση με τις ε, ΠΑ και τις ΜΜΑ, τις μετεγκριτικές μελέτες ασφάλειας, ε, δηλαδή ε, και, ούτως ώστε να, ε, έχουν, να δικαιολογούνται. επίσης το τέλος για τις παραπομπές οι περισσότεροι λένε ότι εκεί δεν είναι αρκετά υψηλό το τέλος αυτό. Πάντως άκουσα πολλά και διάφορα τέλη ε, με βάση του υπολογισμού των κρατών μελών. Από την Ολλανδία είδα διπλάσια νούμερα από αυτά του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι γνώμη έχει η Κομισιόν για τα διάφορα ε, επίπεδα τελών που πληρώνονται και που χρεώνονται από ό,τι φαίνεται από τα διάφορα κράτη-μέλη. Η κυρία Ροτ Μπέρεντ ζητάει τα κράτη-μέλη να ε, καταρτίζουν ε, ε, τιμολόγια πολύ επακριβή σχετικά για λόγους διαφάνειας, για να ξέρουμε πόσο χρεώνουν. Αλλά πώς, έχει να κάνει, πώς συσχετίζεται αυτό με το τέλος κατά αποκοπήν για τις παραπομπές. Αν έχουμε παραπομπή χρεώνεται ένα τέλος. Αν έχουμε διαφορετικά τέλη, θα πρέπει να προσδιοριστεί τι χρεώνεται κάθε φορά. Αλλά δεν ξέρω, μήπως το παρακάνουμε εδώ και δεν έχουμε πολύ διαφάνεια, αλλά έχουμε πάρα πολλά ε, έγγραφα σε σχέση με αυτό που ζητάμε από τα κράτη-μέλη. Γιατί υπάρχουν πολλές διαφορές. Πολλές φορές δεν, οι χώρε με το χαμηλότερο κόστος δεν είναι αυτές που έχουν τους χαμηλότερους μισθούς. Μερικοί έχουν υψηλό κόστος εργασία και χαμηλά τέλη. Οπότε δεν είναι ανάλογο χαμηλό κόστος εργασίας, χαμηλά τέλη. Ας μας το εξηγήσει και αυτό η Κομισιόν. Επίσης, ε, μια ανησυχία που εξέφρασαν αρκετοί ε, ε, συνάδελφοι μέσα από τροπολογίε σχετικά με τα κίνητρα για παραπομπή ε, όταν ας πούμε στέλνουν στην ε, Επιτροπή ε, ΠΡΑΚ για την ε, κάποια προϊόντα που τους απασχολούν λόγω σκανδάλων που υπάρχουν στη χώρα τους και αφορούν την εθνική ασφάλεια. Οι συνάδελφοι ανησυχούν Μήπω ε, ε, το παρακάνουν τα κρατημέλη και φορτώνουν πολύ με παραπομπές στην ΠΡΑΚ, την, φαρμακο... την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνηση. Ε, και εγώ ανησυχώ βέβαια για να μην βρεθούμε σε μια θέση όπου οι χώρες που κάνουν παραπομπές και που θέλουν να κάνουν παραπομπές θα λένε δεν θέλω να κάνω την παραπομπή γιατί θα στοιχήσει πολλά λεφτά, άρα υπονομεύουμε καλύτερα τη δημόσια ασφάλεια. Κυρία Ροτ Μπέραντ, έχει υποβάλει την σχετική τροπολογία 52 και λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να συμβάλλουν στο κόστος των μη κατεπηγουσών παραπομπών. Ε, αυτές, όχι αυτές, ε, δηλαδή όπου υπάρχει σήμα μεγάλο, ε, δηλαδή μεγάλη, μεγάλες ε, επίσης λέει ότι ο συνεισηγητής ή ο εισηγητής δεν πρέπει να είναι από τη χώρα που κάνει την παραπομπή. Εγώ όταν μίλησα με σχετικούς ανθρώπους που κάνουν την δουλειά στη φαρμακοεπαγρύπνηση μου λένε ότι αυτό δεν είναι πρακτικό. Γιατί ισχυρίζονται ότι οι χώρες που κάνουν παραπομπές ή που... Ε, ε, αυτοί έχουν και τα περισσότερα δεδομένα και τις, τις γνώσεις πάνω στο θέμα. Εγώ προτείνω τα κράτη-μέλη που κάνουν παραπομπή να παίρνουν τη μισή αμοιβή δεν ξέρω τι λέει η Κομισιόν, αν γίνεται αυτό, γιατί όταν μίλησα με κάποιους που δουλεύουν στην ΠΡΑΚ μου λένε ότι πιστεύουν ότι μπορούν να σταματήσουν ε, τις υπερβολές στο σύστημα με εσωτερικέ διαδικασίες χωρίς νομοθετικά μέτρα για να σταματήσουν την καταβολή των ε, τελών. Δεν ξέρω η Κομισιόν τι λέει πάνω σε αυτό. Τώρα, ε, κυρώσεις για εταιρείες που λάθος δηλώνονται ως μικρομεσαίες. Κάποιοι υπέβαλαν τροπολογίες που λένε να αυξηθεί το τέλος. Η Κομισιόν λέει 10% να πληρώνουν, αν έκαναν λάθος ε, άλλοι λένε 20, άλλοι 50% παραπάνω η κυρία Γιάννα Κουδάκη λέει να διαγραφεί το τέλος, να μου πει η Κομισιόν και εδώ τι πιστεύει. Στην ε, οδηγία REACH υπάρχει θέμα με αυτές που, δεν, που δηλώνονται λάθος. Βέβαια αυτό είναι ειδική κατηγορία όπου έλαβαν ε, συμβουλές και έκαναν δήλωση με βάση τις τεχνικές δηλώσεις, τις τεχνικές συμβουλές. Ε, ποια είναι σε αυτή την περίπτωση η σωστή κύρωση. Θα πρέπει να έχουμε υψηλότερε κυρώσεις. Υπάρχει ήδη πρόβλημα εδώ. Ε, πρέπει να μας συμβουλεύσουν οι ειδικοί για τη φαρμακοβιομηχανία και τις Έχουμε πολλές τροπολογίες επίσης ε, που είναι από το FPR και το EGA και από τις καινοτόμες εταιρείες και τις εταιρείες γενοσύμων που ζητούν από τον ΕΟΦ να δώσει περισσότερες πληροφορίες ε, σχετικά με το κόστος. Ε, υπάρχει και, υπάρχουν τροπολογίες 78 με 80 εδώ σχετικά με αυτό το θέμα. Θέλω να το δούμε αυτό και να δούμε τι προβλέπει η έκθεση του ΕΟΦ, τι πρέπει να κοινοποιούν δηλαδή και αν ναι, έχουν νόημα αυτές οι τροπολογίες. Ε, επίσης η κυρία Γκροστέτ δεν είναι εδώ, αλλά ίσως η κυρία Γιούζο μπορεί ε, να τη ρωτήσει. Έχει την 102 τροπολογία που λέει ότι μέρος του κόστους για τις παραπομπές φαρμακοεπαγρύπνησης προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ε, τρόπον την 9 μέρη χρηματοδοτείται από τον ενωσιακό προπολογισμό ΕΟΦ. Οπότε δεν έχω καταλάβει ακριβώ ποιο είναι το νόημα τη τροπολογία και πώ εντάσσεται στην όλη επιχειρηματολογία μα εδώ. Γιατί αν έχουμε περάσει από όλε τι λεπτομέρειε κόστο παραπομπή, ποιο θα πληρώνει και πώ θα λειτουργούν αυτά και ξαφνικά λέμε Α, πρέπει να πληρώνονται από τον προπολογισμό τη Ένωση, ε, δεν έχει και πολύ νόημα. Δεν είναι εδώ η κυρία Γκροστέτ εδώ να εξηγήσει τροπολογίε τη, αλλά ίσω μπορούμε να τη ρωτήσουμε. Λοιπόν, είναι πάνω από 100 οι τροπολογίες. Ελπίζω μέσα από διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να καταλάβουμε τι λένε και να καταλήξουμε σε λογικές προτάσεις σχετικά με τα τέλη. Να θυμόμαστε ότι η βασική προτεραιότητα βέβαια εδώ είναι η ασφάλεια των φαρμάκων. Τίποτα από αυτά που θα κάνουμε εδώ δεν πρέπει να υπονομεύσουν την δημόσια ασφάλεια. Και θα πρέπει βέβαια να βρούμε σωστό τρόπο να πληρώνεται το σύστημα που θα φτιάξουμε. Ευχαριστώ. Αρχίζει η συζήτηση τώρα. η Ντάγμα Ροτ που είναι ο σύνδεσμός μας με τον ΕΟΦ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ Ματίας. Έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες. Θέλω να κάνω κάποια σχόλια για να τις διευκρινίσω. Η Λίντα αναφέρθηκε σε μια τροπολογία από τη κύρια Γκροστέτ, την 102. Εγώ δεν την ε, διάβασα όπως, τη, όπως η Λίντα, ότι ε, πρέπει να έρχεται από το κάποιο κρατικό προπολογισμό, από το δημόσιο προπολογισμό, όχι από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Εγώ έτσι τη διάβασα. Αν θεωρούμε ότι η υγεία των ασθενών είναι σημαντική και πρέπει να τους δίνουμε φάρμακα τα οποία εγκρίνονται και σε εθνικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο και αν πούμε ότι η ευθύνη είναι μόνο, βαραίνει μόνο την βιομηχανία τότε δεν, ε, δεν μ' αρέσει. γιατί είναι καθήκον των εθνικών συστημάτων υγείας η συλλογή τέτοιων πληροφοριών. Και δυστυχώς τα κράτη-μέλη δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους τελευταίες δεκαετίες. Δεν είχαμε συνδεδεμένες βάσεις δεδομένων στα κράτη-μέλη και η νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθυστέρησε. Οπότε αυτή η πρόταση ε, θα ε, έδινε κάποιο, θα, θα ευνοούσε την ε, βιομηχανία και είναι σωστό αυτό γιατί η ευθύνη είναι ευθύνη των συστημάτων υγείας κατά την άποψή μου. Τώρα, αυτό με οδηγεί στα άλλα στοιχεία, στα άλλα σημεία της εισηγήτρες. θα δώσουμε κίνητρα για την επαναχρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Και εκεί μπαίνει και το θέμα των εισηγητών συνεισηγητών, τα, το θέμα των τελών, του συνολικού ποσού κλπ. Οι, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ και μήνες ε, με επικεφαλής στις κάτω χώρες και άλλους προσπαθούν να πάρουν περισσότερα λεφτά από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό γιατί θέλουν να αναχρηματοδοτηθούν. Φοβούνται ή αντιλαμβάνονται ότι οι εθνικοί προπολογισμοί ε, μειώνονται. Εγώ καταλαβαίνω αυτές τις, αυτά τα αιτήματα όταν προέρχονται από τη Γερμανία, από, τον Βασιλ, από, το, από τις κάτω κλπ. Αλλά αν δούμε λίγο το παρελθόν, αν δούμε την ποιότητα των εκθέσεων εισηγητών για την προετοιμασία έγκρισης ε, φαρμακευτικών προϊόντων, έτσι, όχι φαρμακοπαγρύπνησης, κανονική νομοθεσία όπου έχει υποβληθεί αίτηση, έχει γίνει έκθεση για την προετοιμασία της διαδικασίας αδειοδότησης. Αν δούμε την ποιότητα αυτών των εκθέσεων, είναι πολύ διαφορετική από χώρα σε χώρα. Και αν κάποιος τους μιλήσει ε, off the record, θα το δέχονται. Κάποιες εκθέσεις είναι πολύ καλές και κάποιες άλλες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθόλου γιατί δεν είναι καλή ποιότητα. Άλλε δε δεν είναι καν σε μια γλώσσα που να μπορούμε να διαβάσουμε. Οπότε γιατί να, γιατί να πληρώνω εγώ για κακή ποιότητα. Έτσι λένε. Γι' αυτό το λόγο τα κράτη-μέλη ε, θέλουν να αναχρηματοδοτήσουν αυτές οι επιτροπές, αυτές τις μελέτες. Οκ, εντάξει, αλλά τουλάχιστον να βελτιωθεί η ποιότητα. Και εκεί θα μπορούσαμε να πιέσουμε την ε, ε, Ένωση Εθνικών Αρχών ε, ε, δεν νομίζω ότι αυτοί θα μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι για τα τέλη για τα οποία θα εισπράττουν. Μετά, μπορεί ένα κρατός μέλος που κάνει παραπομπή να είναι εισηγητής. Έχουμε δει τέτοιες παραπομπές στο παρελθόν. Κοδαΐνη για παράδειγμα, ε, σε σιρόπια για, για βήχα. Γνωρίζουμε ότι αυτή η ουσία έχει παρενέργειες. Όλοι το ξέρουν. Όπως ξέρουμε και τις παρενέργειες των συλληπτικών χαπιών. Ε, ε, γίνεται παραπομπή όμως. Είναι δικαιολογημένη. Το ίδιο και ε, αυτό που ε, έχει δίκιο η Ελίνα που λέει ότι γίνονται παραπομπές για να αποσυστεί το βάρος της ευθύνης από τα κράτη-μέλη. Ε, δεν συμφωνώ με αυτό που προτείνεται για εισηγητές από, το κράτο που κάνει την παραπομπή. Ε, τι σημαίνει αυτό το δεν θα πάρουμε πληροφορίες. Δηλαδή το κράτος μέλος το οποίο παραπέμπει το συγκεκριμένο φάρμακο δεν θα δώσει πληροφορίες αν δεν έχει συγητή. Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Θα ήθελα όμως να του επιβεβαιωθεί αν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή λέμε ότι ένα κράτος μέλος κάνει μια παραπομπή. Δεν μπορεί να είναι η εισηγητής. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος μέλος δεν θα μας δώσει, δεν θα μας παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες, δεν θα συνεργαστεί. Αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Μετά, η, τα τέλη για τις παραπομπές. Εγώ νομίζω ότι ήταν λίγο ψηλά αυτά τα τέλη στην πρόταση. Η Λίντα τα μειώνουν και κάποιοι άλλοι με τροπολογίες τους. Ε, όμως πρέπει να δούμε τι παίρνουν τα κράτη-μέλη. Δεν αμφισβητώ το ότι ένα ποσοστό πρέπει να πηγαίνει στα κράτη-μέλη. Εγώ θέλω όμως να ρωτήσω τι κάνουν με αυτό το ποσοστό και θέλω να τους υποχρεώσω να μου πούν τι έχουν κάνει. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι θα πρέπει οι εκθέσεις να είναι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να είναι σε μια γλώσσα που να είναι χρήσιμη. Αν τα κράτη, οι, εθνικές κρατές των, ε, εθνικές αρχές των κρατών μελών ε, θέλουν έσοδα, και θεωρούν ότι τα άλλα κρατημέλη και ο ΕΟΦ είναι γελάδες οι οποίες πρέπει να αρμέξουν, θα πρέπει να ε, δίνουν και αποτέλεσμα. Και πραγματικά ε, διαφωνώ με πολλές από τις εθνικές αρχές του Διευθυντικού Συμβουλίου, του Management Board. Συμφωνώ με τη Λίντα για τα γενώσιμα. Ε, τα γενώσιμα θα αποτελέσουν, ε, θα αντιπροσωπεύσουν το μεγαλύτερο όγκο παραπομπών στο μέλλον. Ε, δεν υπάρχει δικαιολογία να δώσουμε κάποια επιπλέον προνόμια ε, στα, στα γενώσιμα. Οι τροπολογίες μου πιστεύω ότι είναι δίκες. Ξέρω ότι ο Ευρωπαϊκός Ορισμός Φαρμάκου χρειάζεται ε, τα, χρειάζεται να έχει προπολογισμό. Δεν αφισβητώ το, το τέλος, το ετήσιο τέλος, αλλά θέλω να δω τι δουλειά γίνεται με αυτά τα λεφτά. Η βιβλιογραφία για παράδειγμα. Μετά η κυρία Παρανόβα και άλλοι έχουν υποβάλει τροπολογίες καλές. Πρέπει τα κράτη-μέλη να μην χρεώνουν μια δεύτερη φορά. Δηλαδή ο το μέσο βιομηχανία να πληρώνει σε, για το ευρωπαϊκό σύστημα, αλλά μην χρειάζεται να πληρώνει και η, σε εθνικό επίπεδο ξανά μετά. Αυτό δεν είναι σαφές από το κείμενο. Έχω και κάποιες άλλες τεχνικές τροπολογίες για τη μείωση του διοικητικού βάρους ε, της ε, ε, υπηρεσίας του οργανισμού και επίσης ότι θέλουμε να είναι σαφές για, το, για ποιο λόγο γίνονται οι πληρωμές όταν υπάρχει τέτοιου είδους υποχρέωση. Είναι η τροπολογία 46 για το άρθρο 11. Με τροπολογία 87 επίσης ήθελα να καταστήσω σαφές ότι μπορεί το σύστημα να ξεκινήσει με αιτήσιο κατά αποκοπή τέλος όταν ε, είναι ε, έτοιμο το σύστημα στο ΝΕΟΦ και έξι μήνες μετά. Ε, επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το ε, τέλος θα δίνει ε, αποτέλεσμα γιατί αλλιώς για μικρές επιχειρήσεις θα είναι παραδεκτό. Ευχαριστούμε και τώρα περνάμε <clears throat> στους σκιώδεις. Πιλάρα Γιούζο πρώτα και μετά η συνάδελφος Παρβάνοβα για τους φιλελευθέρους. Πιλάρα Γιούζο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συγχαρητήρια στην συγγήτρια μία ακόμα φορά. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Να ευχαριστήσω και την κυρία Ροτ Μπέρντ για τις εξηγήσει της. Ε, είναι ε, ειδική για αυτά τα θέματα. Η πρόταση έχει ως... Ε, έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες μαζί με την κυρία Γκροστέτ και κυρία Παρβάνοβα γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν στην έκθεση οπωσδήποτε. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διπλές πράξεις τελών και θα πρέπει να γίνει σαφής ε, διαχωρισμός ανάμεσα στις αποκλειστικές αρμοδιότητες του ΟΕΟΦ και στις αρμοδιότητες που, είναι, ε, που βαρύνουν τα κράτη-μέλη. Επίσης, θεωρώ ότι τόσο οι συγητές όσο και οι ε, αναπληρωτές τους θα πρέπει να οι συνεισηγητές θα πρέπει να αμείβονται επαρκώς. Οι υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχουν στην υπηρεσία, στον οργανισμό, θα πρέπει να διευκρινιστούν. Αλλά αν αυτοί κάνουν τη δουλειά, θα πρέπει να αμείβονται κιόλα. Σε ό,τι αφορά τα γενώσιμα, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να χαίρουν μείωση 20% σε ό,τι αφορά το τελικό ποσό του τέλους. Ελπίζω ότι στην συζήτηση που θα γίνει η συγγήτρια μαζί με τους όλους συγγητές θα καταφέρουμε να συζητήσουμε λεπτομερώς όλες αυτές τις τροπολογίες και να καταλήξουμε σε συμφωνίες που θα διευκολύνουν την τελική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ η κυρία Παρβάνοβα και μετά η κυρία Γιάννα Κουδάκη. Παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τη Λίντα και τους συναδέλφους για τη συνεργασία που έχει ήδη ξεκινήσει για το αρχαίο αυτό. Η συνεργασία μας είναι σημαντική για να υπάρξει ένα διαφάνες, σαφές και αποτελεσματικό σύστημα που θα διασφαλίσει την απλή λειτουργία του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνης. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τον ορισμό του κατόχου εξοδότησης της αγοράς. Είναι σαφές να... ότι είναι σημαντικό να υπάρχει σαφής ορισμός ώστε να αποφεύγονται χρεώσεις και τέλη στα κρατημέλη. Ο ορισμός ορίζεται ήδη στην ανακοίνωση της Επιτροπής ε, για τις διαδικασίες εξουσιοδότησης ε, διάθεσης στο εμπόριο. Θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί λοιπόν με αυτό και αυτή εδώ η νομοθεσία. Όσον αφορά τον ορισμό chargeable unit, χρέωσιμη μονάδα, η μικροποιημένη με την πρόταση της Λίντα και βλέπω ότι η Λίντα συμφωνεί για την εξαίρεση των ονομάτων των ιατρικών προϊόντων. Αυτό θα αποτρέψει προβλήματα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με διάφορους τρόπους. Όσον αφορά την αποφυγή διπλής χρέωσης σε εθνικό επίπεδο, μια περιοδική έκθεση παραπομπών ε, και εξελόγηση των μελετών θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ολόκληρης της διαδικασίας ε, αξιολόγησης και να μην χρεώνεται ξεχωριστά σε εθνικό επίπεδο αφού δεν απαιτείται δεύτερη ε, επιστημονική εκτίμηση όσον αφορά τη μείωση του καταποκοπήν ετήσιου τέλου, το προφίλ ασφαλείας της ουσίας, θα πρέπει να αποτελεί το επίκεντρο. Ένα προφίλ ασφαλείας ενός προϊόντος σημαίνει λιγότερη δουλειά για τον οργανισμό. Προτείνω λοιπόν, τη... υποστήριζω την πρόταση της μείωσης του ετήσιου καταποκοπής τέλους ε, για να υπάρχει η αντιμετώπιση, το τέλος θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα ιατρικά προϊόντα ε, στο πλαίσιο της διάταξης και για όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον όσον αφορά τη διαφάνεια για όλες τις ομάδες ε, είναι ένα σημαντικό ζήτημα για να λειτουργούσουν αποτελεσματικά τα τέλη του ΕΟΦ χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια. Πρώτον, όσον αφορά την αξιολόγηση των εκθέσεων της ΕΟΦ, οι εκθέσεις θα πρέπει να παρέχονται στο Συμβούλιο, την Κομισιόν, την ΕΟΚΕ, το Κοινοβούλιο, το Ελεκτικό Συνέδριο και τα κράτη-μέλη. Οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να δημοσιεύονται ως υπό τη μορφή μιας ετήσιας δημόσιας έκθεσης για τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύει η Κομισιόν για το πώς οι δικαιούχοι εξουδοτήσεων της αγοράς θα πρέπει να κάνουν δηλώσεις ε, και για τη μείωση των τελών υπό το άρθρο 75. οποιασδήποτε οι τροποποίησεις στα ποσά θα βασίζονται σε διαφανή σχέση μεταξύ του κόστου του οργανισμού και του κόστου των αξιολογήσεων των εισηγητών. Όλα αυτά διατυπώνται στο άρθρο 9 και βασική της παρακολούθησης του δίκτυου πληθωρισμού στο άρθρο 18 παράγραφος 4. Πιστεύω ότι με τις κοινές μας προσπάθειες και την πρόταση της Κομισιόν που καλωσορίζω θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε βάσει των κριτηρίων ε, απλουστευσής και διαφάνειας την προτείνομενη νομοθετική πράξη. Θα συνεχίσω τη συνεργασία με τη Λίντα και ελπίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ισχυρή θέση που θα υποστηρίξουμε στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γιάννα Κουδάκη. Ευχαριστώ. Α, αυτό απεδείχθη κουτί της Πανδώρας. Συμφωνώ με όσα είπε η Λίντα και τις, ε, σχετικά με τις ερωτήσεις στην Κομισιόν γιατί χρειαζόμαστε διευκρινήσεις όλα αυτά. Ε, κάτι που είπε η Ντάγμαρ μόλις τώρα όμως με έκανε να ξανασκεφτώ. Δηλαδή να μην είναι εισηγητές από το κράτος μέλος της παραπομπής. Συμφώνησα με αυτό όταν είδα την, την ε, τροπολογία, αλλά μετά είπε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να μοιράζονται τις πληροφορίες. Λογικό. Όμως αυτό συνεπάγεται κάποιο κόστος για το κράτος μέλος. Αν δεν υπάρχει κόστος, εντάξει, αλλά αν υπάρχει κόστος πρέπει να το έχουμε κάπως υπόψη μας, διότι μπορεί αυτό να σημαίνει περικοπές κλπ. Τώρα, ποιος ποιες ευθύνες έχει ο παραγωγός, ποιες έχει το κράτος μέλος. Και εδώ είμαι διχόγνωμη. Μου φαίνεται ότι δεν πρέπει να, σταυρώσουμε, να σταυρώνουμε πάντα τη βιομηχανία και να ζητάμε να τα κάνουν όλα αυτοί, αλλά από την άλλη, αν είναι δικά τους τα φάρμακα, πώς μπορώ να περιμένω από τα κράτη-μέλη να τα παρακολουθούν όλα και να είναι υπεύθυνα για όλα. Δεν είμαι σίγουρη. Οπότε εδώ θέλω περισσότερα επιχειρήματα να ακούσω. Τώρα, αυτό για τις αντικσοότητες. Ε, η τροπολογία ήταν ενδιαφέρουσα και είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, ενδιαφέρουσα η προέλευση. Καταλαβαίνω γιατί κατέθεσε την τροπολογία, γιατί όντω οι χώρε αυτέ περνάνε από αντικσοότητες και πάνε να υπερασπιστούν τη βιομηχανία του. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ερωτήσει που χρήζουν απαντήσεων και εύχομαι καλή τύχη στις συμβιβαστικέ τροπολογίε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Τελειώσαμε τον κατάλογο, τον εξαντλήσαμε. Ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις και για τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Αυτό δείχνει πόσο δύσκολη είναι αυτή η πρόταση. Είναι δύσκολες και οι δημόσιες διαβουλεύσεις. Πολλές επικρίσεις ε, συναντάμε στα διάφορα ζητήματα. Βρισκόμαστε λοιπόν στη φάση προβληματισμού και στο Συμβούλιο. Ξεκινώντας από το σύστημα χρηματοδότησης και τα τέλη, στις προτάσεις μας ε, το σύστημα χρηματοδότησης από τα τέλη θεωρήσαμε ότι ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση που ακολουθήσαμε κατά την ε, φάση έγκρισης της ε, νομοθεσίας για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τέλη και παρέχουμε ότι οι υπηρεσίε που παρέχουν αποτελούν αιτία για την καταβολή τελών. Αυτό ευθυγραμμιστεί και με την τρέχουσα κατάσταση όπου χρεώνουμε ετήσια τέλη για συγκεκριμένα προϊόντα και λαμβάνουμε υπόψη και του περιορισμού του προπολογισμού για τι δραστηριότητε που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από αυτόν τον πόρο. Φυσικά τίθεται το σημαντικό ερώτημα του σε... πώς από τα άλλα δημόσια κονδύλια μπορούν να δαπανηθούν για αυτό το σύστημα και ακούμε και επιχειρήματα ότι υπάρχουν και άλλα κόστη που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα κράτη-μέλη, τα νοσοκομεία, γιατροί κτλ. Τώρα γίνονται συζητήσεις για τις χρεώσιμες μονάδες. Οι χρεώσιμες μονάδες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των πληρωμών αλλά θα πρέπει να δούμε από κάθε εταιρεία αλλά πρέπει να δούμε τι αριθμό προϊόντων έχει κάθε εταιρεία στην αγορά. Η παρακολούθηση τώρα και τις ασφάλειες για το κάθε προϊόν. Θεωρούμε λοιπόν ότι το όνομα του ιατρικού προϊόντος πρέπει να παραμείνει κομμάτι αυτού του τουρισμού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ορισμός που υπάρχει στον κανονισμό 2083. Δεν περιλαμβάνει... Δεν πρέπει να παραλαμβάνει και τα παράγωγά του. Ε, θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Τώρα για πρακτικά θέματα αγορά του εδεφορμένου του δικαιούχου πρέπει να θεωρείται ότι ο δικαιούχος δεν είναι η ομάδα όμιλος στον οποίο ανήκει. Είναι σημαντικό ζήτημα αυτό και θέλαμε να το αναφέρουμε. Όσον αφορά τα διάφορα τέλη για τα τέλη παραπομπών για αυτά τα Θεωρούμε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τεράστιε διαδικασίες με πολύ μεγάλο αριθμό φαρμακευτικών προϊόντων με πολύ υψηλότερα κόστη από τα μέσα. Πρέπει να τονίσουμε ότι για τον ορισμό του ποσού του τέλους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κόστος ε, του, που υφίσταται το κράτος Ένα άλλο ζήτημα αφορά τις μεγάλες παραπομπές ε, που υπόκειται σε ψηλότερα τέλη. Πιστεύουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να μεριμνήσουμε για μικρότερες παραπομπές που αφορούν ένα ή δύο δικαιούχους ε, εξοδοτήσεων. Είναι σημαντικό το ποσό για κάθε εταιρεία του τέλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσει οικονομικές δυσκολίες λόγω του ύψους του. Όταν συζητάμε για αυτές τις οικονομικές δυσκολίες, ε, ξέρω ότι σας φαίνεται περίοδο, αλλά είναι σημαντικό ζήτημα. Τέλος, όσον αφορά τις παραπομπές απόψη δημοσίας υγείας, δεν πρέπει να υπάρχουν ε, χρηματικές αποτροπές για τις διαδικασίες φαρμακοϊπαγρύπνησης. Οι παραπομπές λοιπόν δεν πρέπει να κυρώνονται οικονομικά. Ωστόσο, με την αναθεωρημένη νομοθεσία της φαρμακοεπαγρύπνησης τα κράτη-μέλη έχουν λιγότερη διακριτική μεταχείριση για να αποφασίσουν κατά πόσο θα ξεκινήσουν ή όχι οι παραπομπέ. Οι παραπομπέ ουσιαστικά σε πολλέ περιπτώσει επιβάλλονται από την ίδια την νομοθεσία. Επίση, συζητήσαμε με τα πρόεδρο και τα μέλη της ΠΡΑΚΑ και πιστεύουν, όπως είπε και η συγγήτρια, ότι ήδη υπάρχει βελτίωση στην κατάσταση και πιστεύουν ότι μπορούν να διαχειριστούν τη ροή αυτών των παραπομπών. Παρατηρούμε όμως επίσης ότι όλο και περισσότεροι οργανισμοί εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν είναι όπως για την εξουσία τη αγοράς ε, που υπήρχε περιορισμένος αριθμός οργανισμών. Σε αυτήν εδώ την ασκή βλέπουμε ότι όλο και οι οργανισμοί εμφανίζονται και οι και οι για να κάνουν τη δουλειά. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η νομοθεσία αυτή θα εξελιχθεί και θα εφαρμοστεί με καλά αποτελέσματα. Όσον αφορά τα τέλη PCR, επίσης, πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση είναι περιορισμένη. Προτείνονται 90.000 ευρώ. Το υπολογίσαμε βάσει του κόστου του ΕΟΦ και των κρατών Προσπαθήσαμε επίσης να δούμε την εκτίμηση αντικτύπου, ποιο το κόστος για τον ΕΟΦ. Διότι σύμφωνα με τον υπολογισμό μας 30% είναι από τον ΕΟΦ και 70% από τα κράτη-μέλη. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν 600 PCOR περίπου το οποίο σημαίνει ότι ο ΕΟΦ έχει και αλληλένδετες δραστηριότητες με αυτό το τομέα που αυξάνει τις παραπομπές και τις υποθέσεις για το ετήσιο καταποκοπήν τέλος. Δεν πιστεύουμε ότι το χρονοδιάγραμμα πρέπει να βασίζεται στην ημερομηνία απλής λειτουργίας της φαρμακοεπαγρύπνηση. Ο οργανισμό πρέπει να χρηματοδοτήσει τι δραστηριότητε του από τώρα. Η χρηματοδότηση δεν πρέπει να περιορίζεται στη φαρμακοεπαγρύπνηση. Εμείς συζητήσαμε τον οργανισμό και καταλάβουμε ότι αυτό πρέπει να διευκρινιστεί εδώ. Μιλάμε για 1η Ιουλίου ως βέλτιστη ημερομηνία, αλλά θα δούμε τι θα γίνει με τις εξελίξεις της νομοθεσίας. Μετά υπήρχε το πεδίο εφαρμογή των κατευσίδων της πράξεων. Είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο των συζητήσεων μας και στο Συμβούλιο να υπενθυμίσουμε στην Επιτροπή αυτήν ότι το να υπάρχει αυτή η είναι σημαντικό τουλάχιστον για το ετήσιο τέλος διότι το σύστημα τώρα ξεκινάει πολλές παράμετροι επισέρχονται τις οποίες θεωρούμε ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε αρχικά, αλλά θα χρειαστεί να υπάρξει κάποια στιγμή προσαρμογής λόγω του αριθμού των χρεώσιμων μονάδων και των δαπανών που υπολογίζουμε. Τώρα να προσπαθήσω να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις ε, αν με μέγραφες σχόλια, διότι εξαντλείται ο χρόνος. Όσον αφορά το σημαντικό του ερώτημα της ομοιοπαθητικής, προσπαθήσαμε να ελέγξουμε με, την με τον ΕΟΦ πόσες παρενέργειες φαρμάκων οφείλονται σε τέτοια προϊόντα, διότι το κύριο ζήτημα φυσικά είναι η ασφάλεια. Είναι πολύ δύσκολο διότι η σημερινή βάση δεδομένων φαρμακού επαγρύπνησης δεν σχετίζεται με τον τίτλο εξουσιοδότησης ή άλλους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, αυτή τη στιγμή από τις 500 φωτοναθεραπευτικές ουσίες που υπάρχουν στη λίστα, για τις οποίες απαιτούνται PCR, υποβολές PCR, δεν περιλαμβάνεται καμία ομοιοπαθητική ουσία. Όσον αφορά τα γενώσιμα. στη βασική νομοθεσία δεν θέλουμε να υποβάλλεται πίσω άργια συγκεκριμένε αξιολογίε εκτό αν ζητηθεί συγκεκριμένα από το κράτο μέλο. Αυτή τη στιγμή η συμπερίληψη των γεννώσιμων απαιτείται για 10 με 15% των ουσιών τουλάχιστον. Όσον αφορά τι παρενέργειε των προϊόντων που υπόκειται στη βάση δεδομένων τη φαρμακοεπαγρύπνηση, Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν μπορεί να εντοπίσει παρενέργειες συγκεκριμένα για τα γενώσιμα αλλά υπολόγισε ότι από το 2012 παρατηρήθηκαν περίπου 70.000 ε, παρενέργειες που αναφέρθηκαν στο σύστημα φάρμακο επαγρύπνησης Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του αριθμού των ADR και Όσον αφορά την εσφαλμένη δήλωση ε, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δηλώνουν εσφαλμένα κάποια θέματα και εκεί έχουμε το πρόβλημα των ορισμών για τον ΕΟΦ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αυτήν την άσκηση. Επειδή αυτές οι τρεις είναι κυρίως εθνικές, είναι δύσκολο να ορίσουμε το πρόστιμο. Στην πρόθεσή μας προτείνουμε 10% αλλά από ό,τι καταλαβαίνω έχουν γίνει και κάποιες και κάποιες γι' αυτό. η, η αμοιβή συνεισηγητή. Ναι, όντως ε, δεν το λάβουμε υπόψη στην πρότασή μας. Και αυτή η συζήτηση είναι σημαντική στο Συμβούλιο. Είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε. Αλλά το ερώτημα που τίθε είναι πώς θα αυξηθεί αναλογικά αυτό η αμοιβή. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για την κοστολόγηση του προπολογισμού σε εθνικό επίπεδο. Είναι πολύ δύσκολη η σύγκριση μεταξύ κοστολόγησης, τιμολόγησης, τελών, αμοιβών που προτείνονται. Αυτό δείχνει επίσης ε, τι είδους προβλήματα μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε στην επόμενη φάση της άσκησης αυτής κατά το, γενικό, το κανονισμό των γενικών τελών ε, όπου θα χρειαστεί να συνεργαστούμε πιο στενά μεταξύ εθνικών οργανισμών για να καταλάβουμε καλύτερα την τιμολόγηση των διαφόρων ε, δράσεων και ενεργειών. Όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων της ΕΟΦ, όλες αυτές τις δραστηριότητες, διαφάνεια στην τρέχουσα φάση, η ετήσια έκθεση ορίζεται με μια συγκεκριμένη δομή το ερώτημα του πόσο περισσότερα θέλουμε να γνωρίζουμε και σε ποιο επίπεδο είναι δυνατή αυτή η ενημέρωση πρέπει πρώτα απ' όλα να εξετάσουμε πολύ σωστά και να κρίνουμε το διοικητικό φόρτο πριν να αποφασίσουμε την τελική μορφή τέτοιων εκθέσεων. Τι μορφή θα έχουν τελικά και τι μορφή θα έχει τελικά αυτός ο κανονισμός. Θα προσπαθήσουμε να στείλουμε και επιπλέον πληροφορίες, κυρίως νούμερα, ποσοστά, κόστη, απευθείας ε, στην κυρία Συγήτρια. Ευχαριστώ πολύ και τέλος η Λίντα, η Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Το, η συζήτηση για το ποιος πληρώνει τι για την φαρμακοεπαγρύπνηση έχει σχέση με τέλη τα οποία χρειάζονται για συγκεκριμένες εργασίες. Αλλά νομίζω ότι ε, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα χρεώσουμε τέλη για όλες τις εργασίες που γίνονται. Η υποδομή που παρέχει ένα κρατός μέλος δεν είναι δυνατόν ε, να πληρωθεί από αυτά τα τέλη γιατί η υποδομή φαρμακοπαραγνησής κοστίζει εκατομμύρια εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε ε, τα τέλη δεν θα είναι υπερβολικά επουδενή. Και βέβαια το τέλος που σχολιάζουμε εδώ είναι κατά αποκοπήν ενώ ε, τα κόστη διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από επιχείρηση σε επιχείρηση κλπ. Ε, κάποιες επιχειρήσεις ζητούν να υπολογιστεί το πραγματικό κόστος αλλά αυτό θα, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ περίπλοκο. Γιατί γνωρίζουμε ότι θα χρειαζόμασταν τις συμβουλές ε, εμπειρογνωμών που είναι πολύ ακριβές. Ξέρουμε πόσες προσ... Ε, ε, ε, ε, παραπομπές γίνονται και μπορούμε να κατανείμουμε το κόστος, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε πολύ λεπτομερείς ό,τι αφορά τον υπολογισμό του κόστους. Τώρα, ποιος θα έπρεπε να μπορεί να είναι εισηγητής ή συνεισηγητής για τις παραπομπές. Πρέπει να το εξετάσουμε πιο προσεκτικά, να δούμε ποια είναι η σημερινή πρακτική και πώς λειτουργεί το σύστημα τώρα, καταρχήν. Εγώ νομίζω ότι ήδη υπάρχουν κανόνες για το ποιος μπορεί να είναι εισηγητής και ποιος δεν μπορεί να είναι. Θα ήθελα η Κομισιόν να διευκρινίσει το θέμα των μομπραστικών για το οποίο μίλησε ο Πίτερ Λίζε και το θέμα των βοτάνων βέβαια. Μιλάμε για αυτά βέβαια τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην νομοθεσία γιατί πάρα πολλά δεν συμπεριλαμβάνονται. Αν ε, χρειάζεται μια πέα για, τον, για ένα βότανο σκεύασμα, ε, τότε αυτό οφείλεται, ξέρουμε ότι οφείλεται στο γεγονό ότι περιλαμβάνει κάποια δραστική ουσία. Έτσι. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί να ε, μην πληρώνει τέλεια, αφού έχει μια δραστική ουσία η οποία πρέπει να αξιολογηθεί και πρέπει να ερευνηθεί. Ε, δεν νομίζω θα έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις βέβαια. Δεν νομίζω ότι ε, θα υπάρξουν ομοιοθετικά φάρμακα που θα χρειάζονται η περιοδική επικαιροποιημένη έκθεση ασφάλειας, αλλά μπορεί και να υπάρξει αυτή η περίπτωση. Τι να, πώς να το αποκλείσουμε. Μιλάμε όμως έτσι κι αλλιώς για τα προϊόντα τα οποία ε, ε, έχουν ε, υποχρέωση έγκριση, έτσι. Σε πολλά ζητήματα νομίζω μπορούμε να βρούμε λύση και συμβασμό. θα πρέπει να δούμε το θέμα της βάσης δεδομένων του, και του κατά πόσον και πώς θα χρηματοδοτηθεί. Έχει τροπολογία η κυρία Ροτ Μπέρεντς για αυτό το θέμα. θα προσπαθήσω να βρω ε, λύσεις μαζί με τους ηγητές για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα Μακέβαν. Στις 27 σήμερα συζητήσαμε, στις 17 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε την έκθεση και ενδεικτικά λέμε ότι ε, η έκθεση θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση και προχωρούμε στο σημείο 7, την έκθεση της Πιλάρα Ιούζο, η οποία και θα λάβει αμέσως το λόγο. Παρακαλώ κυρία Ιούζο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μιλούμε για την έκθεση για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό. Η πρόταση αυτή έχει πιο απλούς, απλοποιημένους κανόνες για την εμπορία ε, σπόρων από φυτόρια, για τη διατήρηση της παραγωγικότητας ε, και την ποικιλομορφία των δασών και των καλλιεργιών και για να διευκολυνθεί το εμπόριο. Αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν. Ε, ε, καταργεί 12 τομεακές οδηγίες τεχνικού χαρακτήρα και τις αντικαθιστά με ένα οριζόντιο οικονομισμό με 146 άρθρα, 14 παραρτήματα και μας απειλεί με την ε, μελλοντική έκδοση πάνω από 90 πράξεων εκτελεστικών και κατεξιοδότηση από την Κομισιόν. Η πρόταση επίσης διευκρινίζει ότι οποιοδήποτε μη επαγγελματίας, ε, καλλιεργητής, μπορεί να συνεχίσει να ανταλλάσσει σπόρους με άλλους ιδιώτες χωρίς να υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού. Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι νέοι κανόνες λαμβάνουν υπόψη το τύπο του υλικού, τις συνθήκες παραγωγής, το μέγεθος της επιχείρησης κλπ. κλπ. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι ορισμένα είδη, όπως τα, παραδοσιακές για παράδειγμα, ε, θα υπόκεινται μόνο σε κανόνες καταγραφής που δεν θα είναι τόσο αυστηρή όσο ε, ε οι που αφορούν τα άλλα υλικά. Επίσης μειώνεται το διοικητικό άκτος για τις μικροεπιχειρήσεις που μπορούν να εμπορεύονται οποιοδήποτε τύπου εμπορεύματα χωρίς να ε, καταχωρούνται. Οι μικροεπιχειρήσεις επίσης ε, εξαιρούνται από τα τέλη καταχώρησης. Αυτή είναι η πρόταση Κομισιόν. Η θέση μας είναι ότι η ενοποίηση αυτών των 12 τομιακών οδηγιών συνεπάγεται ότι μπαίνουν και υπόκεινται στους κανόνες τομείς πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους ε, και δημιουργούνται στρεβλώσεις και παρεξηγήσεις σε όλους τους συγκεκριμένους κανόνες, σε συγκεκριμένους τομείς. Το κείμενο ε, σε πολλά σημεία είναι πολύ γενικό για τόσο τεχνικά ζητήματα. αλλά αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ε, έχουμε ανεπαρκείς ορισμούς, ε, κάτι που προφανώς θα δημιουργήσει προβλήματα στην εναρμονισμένη εφαρμογή του κανονισμού. Η πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει υπερβολικό αριθμό πράξεων κατά εξοδότηση και εκτελεστικών, πάνω από 90 όπως είπαμε, κάτι που ε, μένουν εκτός της βασικής πρότασης σημαντικά στοιχεία. Στη δική μου έκθεση έχω συμπεριλάβει διάφορους, διάφορες διευκρινήσεις των ορισμών, όπως για παράδειγμα ορισμούς για διάφορα ε, είδη ε, υλικού, και προτείνω την επαναδημιουργία της εμπορικής κατηγορίας, την οποία καταργεί η Κομισιόν. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται επίσημος έλεγχος για, τους, για τα στάνταρ υλικά ε, μετά την θέση του σε εμπορία. Η πρόταση επίσης δεν ορίζει τα είδη που θα πρέπει ε, να πιστοποιηθούν επισήμως, ε, υποχρεωτικά. Ε, παραπέμπει το θέμα σε μια κατεξοδότηση πράξη στο μέλλον. Αυτό θα δημιουργήσει καθυστερήσεις ανεπιθύμητες και θα στρεβλώσει ε, πάρα πολύ ως μέρος Γι' αυτό το λόγο συμπεριλαμβάνω ένα παράρτημα στην εκθεσή μου που καθορίζει ε, θα, που περιγράφει ε, τα είδη που θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρεωτική πιστοποίηση. Η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει και πρόταση, σύμφωνα με την συνήθη νομοθετική διαδικασία, για να, να τροποποιήσει ή να επικαιροποιήσει αυτό το παράδειγμα. Το παράδειγμα αυτό όμως θα πρέπει να υπάρχει. Σε ό,τι αφορά τις ποικιλίε οι οποίες δεν καταχωρούνται, πρέπει να ε, έχουμε μέγιστες προθεσμίες εμπορίας για μικρές ε, περιορισμένες ποσότητες ε, αναπαραγωγικού υλικού. Γιατί αλλιώς θα δημιουργήσουμε μια παράλληλη αγορά ποικιλιών που δεν καταχωρούνται. Σε ό,τι αφορά τα άτομα τα οποία ανήκουν σε οργανώσεις διατήρησης ή συντήρησης, και εμπορεύονται φυτά και σπόρους, η πρόταση της Κομισιόν θέλει να τους εξαιρέσει, όπως είπαμε. Εγώ όμως δεν συμφωνώ με αυτή την θέση, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί μια, ένα παράλληλο δίκτυο φυτικού αναπαραγωγικού υλικού και οι ανταλλαγές μεταξύ ιδιωτών θα πρέπει να περιοριστούν σε μειωμένες ποσότητες, αφού σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται δεδομένο ότι οι ανταλλαγές γενικότερα δεν συνιστούν εμπορική συναλλαγή. Όσο αφορά τι ε, εξαιρέσει από την καταχώρηση στο Μητρό για εξειδικευμένε αγορέ ποικιλίων τοπικού ενδιαφέροντο, είναι απαραίτητο να οριστούν με σαφήνεια οι εν λόγω αγορέ ε, για να αποφύγουμε την αδιάκριτη εφαρμογή της εν λόγω διάταξης. Δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από την καταχώρηση οι μικρές επιχείρησεις δηλαδή επαγγελματίες με λιγότερο από 10 εργαζόμενους και με κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Διότι αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη πλειονότητα του τομέα ε, υλικού. Θα... θα ήταν σαν να εξαιρούμε σχεδόν όλο τον τομέα. Θα πρέπει να καθοριστούν οι μέγιστες ποσότητες που θα μπορούν να επωφελούνται από τις ε, εξαιρέσει αυτέ, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθεί παράλληλο δίκτυο επαγγελματιών που θα διαθέτουν στην αγορά ε, σπόρου ποικιλιών οι οποίε δεν έχουν καταχωρηθεί. Δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια ελέγχων κάθε χρόνο. Η συχνότητά του θα πρέπει να καθορίζεται από τα κράτη-μέλη με βάση τον κίνδυνο ε, παραβίασης ε, των απαιτήσεων. Από την άλλη μεριά η αύξηση των επιθεωρήσεων, ε, δειγματοληψιών ή δοκιμών πρέπει να δικαιολογείται από ανάγκη που προκύπτει από τον έλεγχο και όχι από κάποια ε, τυχαία επιθυμία του επαγγελματία. Άφησα για το τέλος το θέμα που εμένα με απασχολεί περισσότερο. Ίσως δεν είναι το πιο σημαντικό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει ένα νέο μητρό κλόνων. Είναι νέο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κανένα τομέα. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταρριφθεί αυτό το μητρό, να μην το αποδεχτούμε. Ε, πρώτον υπάρχει, γιατί με αυτόν τον τρόπο ε, θα διορθώσουμε ε, ένα ε, λάθος νοοτροπίας. Εγώ δεν ξέρω, δεν, δεν είμαι ειδική για κλόνους, αλλά έχω εργαστεί πάνω από 20 χρόνια καταρχήν στην καταχώρηση επικλειών στη χώρα μου και μετά στην υγειονομική και κλονική ε, επιλογή φυτών. Ξέρω λοιπόν αρκετά πράγματα για αυτό το θέμα. Αυτό που ξέρω όμως ιδιαίτερα ε, ε με βοήθησε να μιλήσω με εμπειρογνώμονες ε, για κλόνους, για κλωνοποίηση φυτών και αυτοί με ενημέρωσαν. Πιστεύω ότι το Μητρό κλόνων θα πρέπει να αποσυρθεί από την πρόταση της Κομισιόν. Και ζητώ από τους άλλους συζητητές να συμφωνήσουν μαζί μου και ε, από όλους τους συναδέλφους γενικότερα. η, η Ένωση Προστασίας ποικιλιών, Φυτικών Ποικιλιών έχει καθορίσει πολύ καλά το τι είναι κλόνη. Όμως η, η νομοθεσία ε, αναφέρεται σε άλλο ορισμό του κλόνου. Οι ενδεχόμενοι διαφορετικοί γενότυποι, λέει που μπορούν να εμφανιστούν στο πλαίσιο μιας ε, ποικιλία και ε, μπορούν να διαχωριστούν με επιλογή. Αυτό δεν είναι, ε, μάλλον δεν είναι δυνατόν να δοθεί σε ένα νομικό κείμενο ένας ορισμός για μια ε, έννοια η οποία έχει οριστεί σε διεθνές επίπεδο. Μπορούμε να συζητήσουμε τι είναι κλόνος στην επικοινία, τι είναι ε, επιλογή κλπ. Αλλά αν κάποιος θέλει να μιλήσει μαζί μου διμερός, ε, πολύ ευχαρίστως, δεν θέλω να ε, επεκταθώ εδώ πέρα. Και μπορώ να μιλήσω και με την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Παύλ Πόκ και μετά η Κορίν Λεπάζου. Παύλ Πόκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω τσέχικα, γι' αυτό βάλτε τα ακουστικά σας. Συμφωνώ και σε κάποιο βαθμό υποστηρίζω την άποψη της εισηγήτριας. Έχω μάλιστα και μια σειρά ερωτήσεων που σχετίζονται με τα ζητήματα αυτά. Ε, μία από αυτές τις ερωτήσεις είναι για ποιο λόγο παρουσιάζεται αυτή η πρόταση σε εποχές όπου με τα θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα στην τρέχουσα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. συζήτησα με πολλούς ενδιαφερόμενους και όλοι μου είπαν το ίδιο. Μου είπαν ότι το σημερινό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σεβαστό παγκοσμίω, θεωρείται εξαιρετικό και πρέπει να διατηρηθεί. Για ποιο λόγο λοιπόν προσπαθούμε να διορθώσουμε κάτι που δεν είναι χαλασμένο. Γιατί να αντικαταστήσουμε 12 τομεακές οδηγίες με μία ενιαία η οποία αποκλείται να καταφέρει να έχει τις ίδιες, τα ίδια καλά αποτελέσματα. Η Κομισιόν προσπαθεί να περιλάβει θέματα όπως το δασικό αναπαραγωγικό υλικό και αυτό είναι εκτός του πιθανού πεδίου εφαρμογής όσον αφορά τους σπόρους και τους σπόρους πουρικής. Πρόκειται για κάτι τελείω διαφορετικό. Είναι διαφορετική τομή. Οποιοδήποτε λοιπόν προσπάθεια να συγχωνευθούν όλα αυτά σε ένα ενιαίο νομοθέτημα είναι καταδικασμένη αυτή εξ αρχή. Ουσιαστικά το κοινό το αμφισβητεί απόλυτα γιατί να καταστρέψουμε κάτι που λειτουργεί για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Σπόρων. Ειλικρινά εγώ δεν έχω απάντηση για αυτό το ερώτημα κοιτώντας τις αναφορές, κοιτώντας τα σχόλια που λαμβάνουμε από το κοινό, βλέπουμε ότι πολλές από αυτές τις αναφορές αφορούν πράγματα που δεν περιλαμβάνονται καθόλου στην πρόταση, όπως η μεταφορά αναπαραγωγικού υλικού, η ανταλλαγή ειδών μεταξύ μη επαγγελματιών, η ε, σάκους γενετικού υλικού ή άλλους σπόρους ε, επιστημονικής έρευνας. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι δεν θέλει να αποδυναμώσει τους σημερινούς κανόνες ε, διότι φοβάται ότι η εικόνα του αναπαραγωγικού υλικού ευρωπαϊκής προέλευσης θα υποβαθμιστεί. Τότε λοιπόν για ποιο λόγο αποδυναμώνεται τους σημερινούς κανόνες. Και αυτό ακριβώς κάνει αυτή εδώ η πρόταση τους αποδυναμώνει τους κανόνες στα περισσότερα κράτη-μέλη. Η απάντηση ίσως βρίσκεται κάπου μέσα στην οδηγία. Ίσως, μέσω τη, ίσως την προτινόμενη ευρωπαϊκή καταχώρηση. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ευρωπαϊκή καταχώρηση. Εάν κάποιος καταχωρήσει τους πόρους του σε εθνικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι ο Εθνικός Οργανισμός αυτόματα θα στείλει στο Ευρωπαϊκό Μητρό τις πληροφορίες. Υπάρχει λοιπόν Ευρωπαϊκό Μητρό από τώρα. Αλλά τι πάμε να φτιάξουμε εδώ τώρα, πάμε να φτιάξουμε ένα εργαλείο ε, διάθεση στο εμπόριο για τις ε, πολυεθνικές. Με αυτόν τον τρόπο θα μπουν στην ευρωπαϊκή αγορά από την πίσω πόρτα και δεν μπορώ καν να φανταστώ ποια θα είναι η τελική έκβαση όλων αυτών. ξεφορτωθήκαμε την άκτα ως μέσο το οποίο θα παραβίαζε κατάφορα τα δικαιώματα των πολιτών και τώρα αφού πετύχαμε αυτό εμφανίστηκε αυτή εδώ η πρόταση και πιστεύω ότι περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία τα οποία πραγματικά θα μπορούσαν να πλήξουν την αγορά και τη το βιομηχανία των σπόρων στην Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά τις κατεξουδότηση πράξεις, η Κομισιόν υποτίθεται ότι προβλέπει 90 επιπλέον κατεξουδότηση πράξεις. Θεέ μου, πρέπει να ψηφίσουμε μια τέτοια πρόταση που δίνει επιταγή λευκό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα... Εγκρίνουμε δηλαδή εμείς κάτι και λέμε στην Κομισιόν εσείς θα ορίσετε τις λεπτομέρειες. Είναι εντελώς παράλογο. Είναι κάτι απαράδεκτο. Τώρα όσον αφορά τις μικροεπιχειρήσεις. Έθεσε το θέμα πολύ σωστά η συγκήτρια. Αναφέραμε την πρόταση ως έχει. Αυτές οι εταιρείες εξειδικευμένων αγορών εύκολα θα μπορούσαν να προμηθεύουν ολόκληρη την αγορά της δικής μου χώρας όχι μόνο με μικρά πακετά σπόρων για τους κυπουρούς αλλά και με σπόρους για δημητριακά. Διότι ο ορισμός δεν έχει κανένα νόημα. Θα μπορούσε να καλύπτει σχεδόν οποιαδήποτε εταιρεία σπόρων. Ας επιστρέψουμε λοιπόν σε αυτά που ορίσαμε στην κοινή γεωργική πολιτική. Ορίσαμε τους μικρούς αγρότες στην κοινή γεωργική πολιτική. Ας επιστρέψουμε σε αυτό τον ορισμό. Το άρθρο 36 χρειάζεται μεγαλύτερη αναδιατύπωση, περισσότερη διατύπωση, διότι υπό την τρέχουσα μορφή του βλάπτει τους πάντες. Εάν αυτή η πρόταση θέλει να ασχοληθεί με τη σημερινή, όχι ακριβώς νόμιμη ή παράνομη ουσιαστικά κατάσταση όπου υπάρχει σκιώδης αγορά σε κάποια κράτη-μέλη για τους σπόρους, η πρόταση πρέπει να έχει τελείως διαφορετική μορφή. Έτσι όπως έχει σήμερα, η πρόταση αυτή δεν επιλύει τίποτα. Όσον αφορά έναν κατά την άποψή μου το βασικό ερώτημα είναι το εξή. Ποιο ήταν το πρόβλημα. Τι θεωρήθηκε προβληματικό από τα κράτη-μέλη και θεωρείται ότι πρέπει να επιληθεί από ένα κανονισμό στο τέτοιο βαθμό. Κανείς δεν μου εξήγησε ποτέ ποιο είναι αυτό που η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θεωρούν ως πρόβλημα τέτοιο που θα πρέπει να καταστρέψουμε το σημερινό καθεστώς μέσω μιας τέτοιας νομοθεσία. Και η άλλη μου ερώτηση είναι τι προσθέμενη αξία προσφέρει ο κανονισμός αυτός. Εγώ δεν βλέπω να προσθέτει τίποτα. Θα απλοποιήσει κάτι. Ίσα ίσα θα κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι επιζήμιο για όλους. Έχω λοιπόν πολύ σοβαρές επιφυλάξεις. Και υποστηρίζω την εισηγήτρια στην ιδέα ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής μέσω τροπολογιών, αλλά δεδομένου του χρονοδιαγράμματος που έχουμε στη διάθεσή μας, ε, αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο. Και πρέπει να πω ότι θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά το κατά πόσο θα υποβάλω μια τροπολογία να απορριφθεί η όλη πρόταση και να επανασταλεί στην Κομισιόν και να επιστραφεί στην Κομισιόν γιατί δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο σε αυτό τη φάση πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Good. Σαφέστατος είσαστε. Ε, συνεχίζουμε με την Κορίν Λεπάζ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Ισηγητρή για αυτήν την έκθεση. Το θέμα είναι εξαιρετικό, εξαιρετικά σημαντικό γιατί οι σπόρ βρίσκονται στην ε, βάση της ε, ε, διατροφικής και της αυτονομίας μας, όμως πρέπει να διατηρήσουμε την ύπαρξη και την ποικιλία σπόρων που είναι προσαρμοσμένοι στις καιρικές συνθήκες και στις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής. Είναι λοιπόν και ευληματικό θέμα. Οι πολίτες μας καταλαβαίνουν τι παίζεται. Αυτή η σπορή είναι σε μεγάλο βαθμό δημόσιο αγαθό και η ανταλλαγή τους ε, γίνεται και σε μη εμπορικά πλαίσια πολλές φορές και θα πρέπει να παραμείνει εκεί. Η πρόταση κομισιών είναι ενδιαφέρουσα. Χρειάζονται κανόνες που να προσαρμόζονται. Για παράδειγμα, βιολογικοί σπόροι ε, θα πρέπει να υπόκειται σε διαφορετικούς κανόνες από τους ε, βιομηχανικούς πόρους. Η Κομισιόν γνωρίζει αυτές ε, τις ανάγκες και γι' αυτό το λόγο έχει κανόνες για ετερογενή υλικά και προβλέπει μάλιστα και εξαιρέσεις. Τι συγχαίρω αυτό. Επίσης κάνει μια χειρονομία καλή θέλησης για τους κυπουρούς, ε, ανθρώπους που παράγουν ε, σπόρους για δική τους χρήση. Είναι σημαντική η, σημαντικό οι ανταλλαγές ανάμεσα σε γεωργούς να αναγνωρίζονται όπως το κάνει το κείμενο. Χρειάζεται όμως οι ορισμοί να γίνουν πιο σαφείς. Ιδιαίτερα ο ορισμός του ετερογενούς υλικού που δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μείγματα ούτε να έχει λάβει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η ε, ε, ζητά την κατάρριση των κλώνων. Συμφωνώ με αυτή την πρόταση οι μικροί αγρότες, γεωργοί, οι οποίοι ε, παράγουν μικρέ ποσότητε σπόρων δεν θα πρέπει να θεωρούνται ω επιχειρηματίε. Γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να δοθεί καλύτερο ορισμό των επιχειρηματιών. Οι ανταλλαγή μικρών ποσοτήτων θα πρέπει να εξαιρεθεί ε, να εξαιρεθούν τις, ε, α, α, νομοθεσίες, ιδιαίτερα για τις εξειδικευμένες αγορές, σε ό,τι διαφορά τις μικροεπιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις. Ε, τα κριτήρια των 10 εργαζομένων και των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά θα πρέπει να δίνεται εξαίρεση για τις ενώσεις, των οποίων βασικός στόχος είναι η διατήρηση, γιατί εκεί χρειάζονται περισσότεροι εργαζόμενοι. Οπότε ε, το κριτήριο 10 εργαζομένων δεν μπορεί να εφαρμοστεί για αυτές. Σε ό,τι αφορά ε, τα φυτά τα οποία υπόκειται σε ε, ανοιχτή αναπαραγωγή δεν μπορούν να συμπεριληφθούν. Είναι κάτι διαφορετικό, ενώ οι έλεγχοι και οι καταχωρήσεις θα πρέπει να γίνονται από δημόσιους φορείς και να μην υπόκειται σε αυτό έλεγχο. Γιατί οι επιχείρησεις αυτές δεν πρόκειται να το κάνουν ή τουλάχιστον όχι μικρές μικρέ επιχειρήσει δεν μπορούσαν να το κάνουν. Θα είχαμε μόνο πολύ μεγάλε επιχειρήσει που θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το έλεγχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Χάση. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια που διευκρίνηση τις απόψεις της και για το σχέδιο έκθεσης που μας ε, παρουσίασε. Μπορώ να συμφωνήσω σε ορισμένα ζητήματα με την εισηγήτρια και σε κάποια άλλα ζητήματα δυστυχώς δεν μπορώ να συμφωνήσω. Η εισηγήτρια κυρία Γιούσα πολύ σωστά θέτει σε αμφισβήτηση την ανάγκη αυτής της πρότασης του συνολό τη. διότι η τρέχουσα νομοθεσία δεν είναι παλιά δεν έχει εκφραστεί κάποια δυσαρέσκεια σοβαρή και ουσιαστικά τα κράτη-μέλη δεν έχουν ζητήσει τέτοιου είδους νομοθεσία. Για τους πρασίνους λοιπόν πιστεύω ότι οι πράσινοι πιστεύω ότι θα εγκρίνουν την απόρριψή της στο σύνολό της. Επίσης συμφωνώ με το ότι πολλά πράγματα στην πρόταση της Κομισιόν να αποκείται σε κατεξοδότηση πράξης υπερβολικά πολλά. Τόσες πολλές κατεξοδότητες πράξεις πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτές. Υπάρχουν όμως και κάποια ζητήματα ε, για τα οποία πράσινα έχουν διαφορετική προσέγγιση από την εισηγήτρια. Το πιο σημαντικό σχετίζεται με την ανησυχία μας για τη βιοπικιλότητα. Για μας λοιπόν, βασική ανησυχία όσον αφορά αυτή την νομοθεσία είναι η προβλέψη της ε, γεωργικής, ε, η προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας αλλά και η προστασία των δικαιωματών των γεωργών να κάνουν ενημερωμένες επιλογές και ελεύθερες επιλογές. Η πρόταση της εισηγήτριας ε, από την άποψη των μικρών φορέων περιορίζει την πρόταση ακόμη περισσότερο σε σχέση με την Κομισιόν δεν μπορώ να συμφωνήσω. Γνωρίζουμε ήδη πολλά για τη σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας. Όχι μόνο στην αγρία φύση, αλλά και στη γεωργία. Η ποικιλία των καλλιεργειών μας ε, κατά κάποιον τρόπο αποτελεί μια ασφάλεια, μια ασφάλιση για μελλοντικές αλλαγές ε, που δεν μπορούμε να προβλέψουμε σήμερα στο σύνολό τους. Κανείς λοιπόν δεν γνωρίζει τι ιδιότητες ε, παραδοσιακές ποικιλίε και τι ιδιότητες θα χρειαστεί να έχουν ετερογενείς ποικιλίε και παραδοσιακές καλλιέργειες στο μέλλον για την ανάπτυξη ποικιλιών που θα χρειαστούμε όταν θα έχει προχωρήσει η κλιματική αλλαγή ή όταν εμφανιστούν ε, νέες ε, καταστροφικές ασθένειες που θα ε, εξαφανίσουν ορισμένες ποικιλίε όπως συνέβη με κάποιες ποικιλίες μπανάνας. Δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει για τις λεπτομέρειες που πρέπει να χαρακτούν κάποια όρια κτλ. Αλλά Αυτό που θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι οι φορείς εκείνοι που προσπαθούν να προστατέψουν ε, και να διατηρήσουν ζωντανές παραδοσιακές ποικιλίε και τη γεωργική βιοποικιλότητα στο συνολό τη. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τα λαχανικά και τα δασικά είδη πρέπει να προστατευτούν. Σε γενικές γράμμες, ε, οι προτάσεις της κυρίας Αγιούσου για τα όρια, για το που θα πρέπει να εφαρμόσετε αυστηρότερο σύστημα και που όχι, εμείς ε, μάλλον έχουμε την αντίθετη άποψη. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα για εμάς είναι η διαφάνεια. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα διάφορα υλικά, τα επίμαχα υλικά, να μην αποτελούν το αντικείμενο λαθρεμπορίου. όλα τα επίμαχα υλικά και τα γενετικώς τροποποιημένα. Θέλουμε να είναι πολύ διαφανές το καθεστώς για αυτά. Επίσης πιστεύουμε ότι η παραδοσιακή ανταλλαγή μεταξύ γεωργών ε, στο πλαίσιο των σπόρων, ανταλλαγή σπόρων, θα πρέπει να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογή του παρόντο κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλους κοιόδης. Τώρα είναι η Λίντα Μακάβαν. Θα αντικαταστήσετε εσείς τον Χανί. Ευχαριστώ. Ναι, εξ ονόματος του Τζιμ ήθελα να μιλήσω, ο οποίος ευχαριστεί την κυρία Γιούζο, όπως πάντα, για τη δουλειά της στην Καλή. Δεν είναι εδώ για να απαντήσει στον κύριο Ποκ, ο οποίος έκανε χρήσιμες παρατηρήσεις. Μπορώ εγώ να απαντήσω για λογαριασμό του. Ε, βέβαια θα ακούσουμε και τι θα πει και εκείνος Νομίζω ότι η πρόταση είναι σοβαρή και πρέπει να τη συζητήσουμε και θα πρέπει να δούμε προσεκτικά τις προτάσεις της Κομισιόν. Τώρα, ο, η υπόθεση του Τζιμ. Υπάρχουν θετικά βήματα στην πρόταση της Κομισιόν, επιλογή, ε, κατα, καταχώρηση σε επίπεδο ενωσιακό θα μειώσει κόστος ε, κατα, ε, ε κόστος, χρόνο, αλλά θα πρέπει να γίνει σωστά η διαδικασία αυτή και δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, γιατί όλα αυτά είναι ασαφή, θολά, δεν έχουμε λεπτομέρειες. Θέλουμε να δούμε ε, βασικούς κανονισμούς που θα ρυθμίζουν ε, τα θέματα των παραγωγών για διασφάλιση ποιότητας και πάλι δεν έχουμε δει σχετικές ε, προτάσεις. Πολλές εκτελεστικές και κατεξουσιοδότηση πράξεις προβλέπονται, τώρα λείπουν. Πολλές φορές η χρήση τους δεν είναι αιτιολογημένη, θεωρούμε ότι δεν χρειάζονται. Ε, θα πρέπει να δούμε εάν ευθυγραμμίζονται με το πεδίο εφαρμογής ε, των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Επίσης ε, θα μπορεί έτσι να θεσπίζει κατεξουσιοδότηση πράξης επαορίστο και αυτό πάντοτε χτυπάει ένα καμπανάκι προειδοποίησης γιατί πρέπει να γίνει εδώ. Τώρα για την απλούστευση, μεγάλη λέξη αυτή, όλοι ε, ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση πρέπει να είμαστε υπέρ της απλούστευσης, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ είναι μία λέξη χωρίς να στηρίζεται από την πρόταση. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και ανησυχώ ιδιαίτερα για τα προκυπευτικά που πολλούν ε, μικρή παραγωγή. Και θέλω να δώσω μια προσωπική άποψη. Εγώ είμαι αυτή, όχι ο Τζιμ πρόσφατα ήρθαν να μου κάνουν λόμπι μια εταιρεία σπόρων από το Ηνωμένο Βασίλειο και μιλούσαν και για ένα κυπευτικό που το φυτεύω και το έχω και εγώ. Λέγεται Sutherland Kale. Ε, είναι στο βορρά του Sutherland. Διαφέρει από άλλες ποικιλίε γιατί ε, δεν θα γίνει εμπορική χρήση του. Ε, επειδή είναι όπως λέμε σε ανεμοδαρμένα ύψη στο βορρά και αντέχει στον άνεμο. Ε, εγώ έχω ε, ένα μικρό αριθμό φυτών που θεωρείται μεγάλος για τα, τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, τα δεδομένα τους, αλλά όχι για εδώ. όσοι εμπορεύονται θα έλεγαν ότι είναι περίπου ε, ε, πουλάνε περίπου 600 κουτάκια το χρόνο, δηλαδή δύο χρόνια θα πρέπει να πουλάνε για να μπορούν να πληρώσουν τα τέλη ε, ή να έχουν, προ, για να έχουν και για να έχουν κέρδη θα πρέπει να περάσουν καμιά δεκαριά χρόνια. είναι λίγοι αυτοί που το καλλιεργούν γιατί από ό,τι φαίνεται το κρατούν, κρατούν το σπόρο για κάποια χρόνια και δεν το καλλιεργούν κάθε χρόνο. Γιατί αυτά τα είδη θα πρέπει να υπόκεινται σε νέους κανονισμούς. Δεν εντοπίζομαι ωφέλη από όλο αυτό το εγχείρημα. Ε, η Κομισιόν θα πρέπει να ενημερώσει το Συμβούλιο ότι έχει λάβει υπόψη αυτές τις ανησυχίες ε, που αφορούν τα θέματα γενικότερα και, όπως και τις προϋποθέσεις για καταχώρηση και θέλουμε να μας πείτε Πώς θεωρείτε ότι οι τροπολογίες αυτές μπορούν να λάβουν χώρα πριν κληθούμε να ψηφίσουμε την πρόταση και αν και το επανεξετάζουν το θέμα σημαίνει ότι επανεξετάζουν τη λογική ολόκληρη της πρότασης ή μόνο το άρθρο 50. Ε, τα κριτήρια συμπερίληψης των ειδών στο παράρτημα 1 για προϋποθέσεις ε, καταχώρησης κλπ. Αυτό σημαίνει ότι ε, όλα τα είδη θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Ε, πολύ αντιφατικά όλα αυτά. Η τροπολογία 21 της κυρίας Σαγιούζο ε, αναφέρεται σε αναθεωρήσεις. Βοηθάει, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να τροποποιήσουμε μόνο το άρθρο 11 και να ε, εξαιρέσουμε όλα τα βασικά. Ε, υπάρχουν λήψεις, δεν προβλέπονται νέες διατάξεις που, ή υπάρχουν διατάξεις που θα επηρεάσουν υπέρμετρα και δεν ε, στηρίζονται οι προτάσεις σε πραγματικές αναλλακτικές και ε, αντικειμενική δουλειά. Επίσης ε, επηρεάζονται οι μικρές αγορές και, και καλλιέργειες ειδική χρήσης ή πωλήσει σπόρων σε ε, γεωργούς βιολογικής γεωργίας ή μικρούς καλλιεργητές. Ε, όλα αυτά τα είχαμε και έχουν αφαιρέσει. Είχαμε ένα σύστημα λειτουργικό και το καταστρέφουμε. Γιατί προτείνει η Κομισιόν ε, να ε, επεκταθούν οι λειτουργίες ε, του γραφείου σε νέους τομείς χωρίς να στηρίζεται αυτό από, από χρώσεις ενδείξεις. Γιατί θα ήταν χρήσιμο κάτι τέτοιο εκτός από το να επιβάλλει περισσότερους ελέγχους. Και γιατί εμείς να, να συμφωνήσουμε με κάτι τέτοιο. Ποιο το όφελος. Τέλος, ε, ο εξυγχρονισμός, ε, η ενημέρωση του κειμένου. Υπάρχουν πολλά άρθρα, το 36 για τις εξειδικευμένες αγορές, τις εξαιρέσεις. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι τόσο θολό και μακροσκελές. Μπορεί να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Ε, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι η προσπάθεια που πρέπει να κάνουν οι υπεύθυνοι νομοθέτες. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκέρλινγκ και τώρα η Λίντα Μακέβαν και ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το δεύτερο νομοθέτημα σήμερα όπου προσπαθούμε να συγχωνεύσουμε τεράστια ποσότητα νόμων σε έναν για να έχουμε απλούστευση αλλά ταυτόχρονα φαίνεται η διαδικασία να είναι εξαιρετικά περιπλοκή και να καταλήγει σε πολλές κατευσίδωτες πράξεις. Φαίνεται δηλαδή απλούστερο αλλά δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μας το σύστημα των κατεξοδοτών της πράξεων δεν λειτουργεί καλά για να επιλύουμε προβλήματα, διότι καλούμαστε να εγκρίνουμε, να απορρίψουμε τροπολογίες. Ε, τις προλήσεις είχαμε πρόβλημα με τα ωραία των πιλότων. Μπορούμε να δεχτούμε ή να απορρίψουμε τις τροπολογίες χωρίς να τις τροποποιήσουμε. Αυτό το ζήτημα όπου προσπαθεί να ενοποιήσει τα πάντα η Κομισιόν ε, και για ποιο όφελος, όπως είπε η κυρία Γκέρλινγκ. Δηλαδή, το πρώτο ερώτημα είναι τι πρόβλημα είναι αυτό που θέλουμε να επιλύσουμε και πώς. Εάν δεν έχει αναφερθεί ως πρόβλημα, γιατί να το λύσουμε. Το ίδιο έγινε και με την υγεία των ζώων. Ξαναγράψαμε... Γιατί να ξαναγράψουμε νόμους που λειτουργούν. Με ανησυχεί και η χρονική στιγμή που παρουσιάζονται αυτές τι προτάσεις. Στο τέλος της θετίας ε, δεν πρόκειται να προλάβουμε να ασχοληθούμε με αυτές σωστά. Θεωρώ ότι η Κομισιόν πρέπει να έχει συνείδηση ότι το να υποβάλει προτάσει τέτοιε στο τέλο τη θητεία, ε, όταν χρειάστηκαν χρόνια για να βγουν από την Επιτροπή, δεν μπορείτε να αναμένετε από το Κοινοβούλιο να βρει λύσει σε πέντε λεπτά, όταν εσεί χρειαστήκατε 4-5 χρόνια για να γράψετε την νομοθεσία. Ασκεί υπερβολική πίεση σε εμά. Ε, εγώ ασχολούμαι με τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Κάνει δύο χρόνια να τη γράψει η Κομισιόν και μετά εμένα μου λένε βιαστείτε. Ε, δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό άλλο αυτή η πίεση και την ταχύτητα. Με ενδιαφέρει το, αυτό που ακούσαμε για καλοπιστικές ποικιλίε και το ζήτημα των διακοσμητικών αυτών φυτών ε, τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από καλλιεργητές ότι θα κοστίσει αυτό πολλά χρήματα με πολύ μικρό κέρδος και η Γκέρλινγκ ε, είπε ότι η Κομισιόν να το αποσύρει αυτό. Θέλω... Για να το πω καθαρά στην Κομισιόν, αυτή θα εξελιχθεί σε άλλη μια ιστορία κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλη την Ευρώπη. Κάθε εφημερίδα και συνάδελφοί μου από την Αυστρία μου νεύουν εδώ. Πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά πριν ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Τι κερδίζουμε από όλο αυτό. Τι προσπαθείτε να επιτύχετε. Νομίζω ότι όλα αυτά δεν βασίστηκαν σε πολλές ε, σε μελέτη των επιπτώσεων επαρκή. Και άκουσα ότι θα υποβληθεί η τροπολογία για απόρριψη της προθέσης και εμείς το ίδιο θα κάνουμε. Μάλλον θα υπάρξει συνένεση, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να καθόμαστε εδώ πέντε μήνες πριν τις εκλογές με ένα τεράστιο νομοθέτημα σαν αυτό προσπαθώντας να βγάλουμε άκρη. Θα πρέπει να εξεταστεί σε περισσότερο χρόνο και σωστά αργότερα. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, είμαι σκιώδης για την ομάδα μας στην Επιτροπή Γεωργίας και χθες ακούσαμε ε, την έκθεση Σιλβέστρης. Είχαμε και μία κρόαση εμπειρογνωμόνων και θέτω το ίδιο ερώτημα κι εγώ γιατί χρειάζεται αυτή η νομοθεσία. Κανένας ε, σύνεδρος δεν ε, το υπεράσπισε. Ακούσαμε ότι η Ευρώπη στο θέμα των σπόρων, των, ε, του αναπαραγωγικού υλικού, έχει εξαιρετική νομοθεσία. Οι 12 οδηγίες ήταν μέχρι τώρα εξαιρετικές. Δεν ξέρω αν υπήρχε λάθος μετάφραση όταν μίλησε ο Πάβελ Ποκ που είπε ότι τώρα πρέπει να συμπτυχθούν σε κανονισμό. Εδώ είμαστε περήφανοι γιατί το εθνικό περιθώριο ελιγμών που υπήρχε εμείς το περιορίζουμε. Και ο τίτλος της δέσμης είναι πιο έξυπνοι κανόνες για πιο ασφαλή τρόφιμα. Εδώ μιλάμε δασικά, ζωικά, φυτικά και το πεδίο εφαρμογής των πρώην 12 οδηγιών κάλυπταν 250 ποικιλίε και τώρα πάμε να καλύψουμε 300.000, δηλαδή όλο το φυτικό υλικό που υπάρχει σε αυτό το πλανήτη. Αυτό το ρώτησα και χθε και δεν μου το απάντησαν. Ε, ακούσαμε πολλές ενστάσεις σήμερα, εγώ θα μπορούσα να συμφωνήσω με τις προτάσεις του εισηγητή, γιατί νομίζω ότι πρέπει να το ξαναστείλω με το κείμενο στην Κομισιόν. Δεν έχουμε λόγο να καταθέσουμε τόσο πολλές τροπολογίες μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, μα δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα προλάβουμε και ότι θα γίνει καλό το νομοθέτημα. Ε, ποιος θα ωφεληθεί από όλα αυτά. Υποθέτομαι αλλά αυτό δεν είναι προς όφελος της βιοποικιλότητας. Χθες ακούσαμε κάτι γιατί μιλάμε για, για φυτά και φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και γιατί πρέπει να πιστοποιείται. Ε, γιατί αλλιώς θα αγοράζαμε γουρούνι στο σακί, όπως λέμε, και δεν θα ξέραμε τι φυτά θα είχαμε τον επόμενο χρόνο και αυτά τα οποία μας υποβάλλει η Κομισιόν είναι γουρούνι στο σακί. Αγοράζουμε κάτι που λόγω των πολλών κατεξουσιοδότηση πράξεων δεν ξέρουμε τι ακριβώς σπόρος θα είναι, πώς θα χρησιμοποιηθεί κλπ. Από τη δική μου την πλευρά, αν δεν υπάρξει ριζική αλλαγή, δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να συμφωνήσω δεν θα ωφελήσει το τμήμα το τομέα των σπόρων και του αναπαραγωγικού υλικού ούτε τους καταναλωτές ούτε θα ωφελήσει τη βιοπικιλότητα ενώ νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και ούτε θα ωφελήσει το Κοινοβούλιο τη στιγμή που συζητείτε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ την κυρία Κάντενμπαχ. Συνοψίζομαι χρειάζεται περισσότερη εργασία και να δούμε τι συνέχεια θα δοθεί. Εγώ είχα προβλήματα με αυτή την πρόταση με την Κομισιόν. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι η αναπομπή. Αλλά η Κομισιόν έχει το λόγο για να μας πει. Θέλει κανείς να μιλήσει. Αν όχι, τότε η συγγήτρια θα λάβει το λόγο. Θέλει. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κάποιες σκέψεις σχετικά με το σκεπτικό του κανονισμού. Το όλο εγχείρημα άρχισε με μια αξιολόγηση του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού και το σύστημα που το διέπει, όπως ζήτησαν κάποια κράτη-μέλη. Και η αξιολόγηση ε, κατέδειξε κάποια θέματα που θα έπρεπε να τα πιάσουμε μέσα από νέο νομοθετικό πλαίσιο. Θα απαριθμίσω κάποια προβλήματα. Ε, συνθετότητα, κατακαιρματισμός του τωρινού νομοθετικού συστήματος με 12 οδηγίες που δεν είναι όλες σχετικά καινούριε. Υπάρχουν οδηγίες από το 1966 και το 1970. Ε, δύο οδηγίες μόνο είναι πιο πρόσφατες. Και ε, αναπτύσσονταν επί 30 χρόνια. Οι 12 οδηγίε λοιπόν λάμπαναν υπόψη διαφορετικά τεχνικά υπόβαθρα και διαφορετικές προσεγγίσεις. Πράγμα που οδήγησε όπως σας είπα σε έναν κατακαιρματισμό του συστήματος. Επίσης υπήρχε ανάγκη ευθυγράμμισης των 12 οδηγιών με, το, με ένα σύστημα που προέβλεπε η συνθήκη της Λισαβόνας και χρειάστηκε βελτίωση τότε. Ε, αυτό εντοπίστηκε στις διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις και σε ό,τι αφορά την απλούστευση, την ε, καλύτερη λειτουργία των ε, εμπόρων, την βελτίωση των γενετικών πόρων και το επίπεδο εναρμόνισης μεταξύ κρατών μελών. Και η ενοποιημένη προσέγγιση που υιοθετήθηκε επιβεβαιώθηκε κατά την προετοιμασία του προγράμματος δράσης και κατά τις διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό τώρα ε, συζητάμε αυτή την πρόταση η οποία διατηρεί τις βασικές αρχές της παρούσας ισχύουσας ε, νομοθεσίας, δηλαδή καταχώρησης των ποικιλιών και της πιστοποίησης πριν από την εμπορία, αλλά θέλει ισορροπημένη προσέγγιση ανάμεσα στην ε, παροχή ενημερωμένης ε, επιλογής όλων αυτών που έχουν ε, παραγωγικό υλικό, αναπαραγωγικό υλικό και αυτών που το εμπορεύονται, το παράγουν, το εμπορεύονται και ε, αυτών που είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση των φυτικών αναπαραγωγικών πόρων. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι τωρινές 12 οδηγίες που είναι σε ισχύ ή μάλλον το παρόν πλαίσιο στηρίζεται σε 12 οδηγίες και 90 δευτερογενείς πράξεις. Οι εκτελεστικές και η κατεξουσιοδότηση πράξη προβλέπονται στις νέες προτάσεις αποτελούν ε, ένα ε, αν θέλετε, ε, μια βασική απογραφή, έναν κατάλογο ε, νομοθετημάτων, που συνολικά θα είναι περίπου 30. Επίσης, υπάρχουν κάποια θέματα που αφορούν κάποιες νέες αντιλήψεις που εισάγονται από τις νέες προτάσεις. Θα ήθελα ειδικότερα να αναφερθώ στις εξειδικευμένες αγορές για να πω ότι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δημιουργήσει ευέλικτο σύστημα που επιτρέπει την εμπορία μεγάλης ποικιλία υλικού πράγμα σημαντικό για πολλούς πολίτες αλλά και για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση των φυτικών γενετικών πόρων. Θέλουμε να συζητήσουμε εναλλακτικά κριτήρια για τις εξειδικευμένες αγορές, όχι με βάση το μέγεθος της επιχείρησης δηλαδή, αλλά με βάση ε, την μικρή αλυσίδα ε, εφοδιασμού, ε, μικρές επιχειρήσεις κλπ. Ένα άλλο θέμα αφορά το ετερογενές υλικό και βλέπουμε ότι αυτού του τύπου το υλικό είναι επίσης σημαντικό ιδιαίτερα για τη βιολογική γεωργία και την υψηλή ανθεκτικότητα σε κάποιες ασθένειες και ζυζάνια. Πρέπει να υπάρξουν ορισμοί εδώ. Ήδη συστήσαμε ομάδα εργασίας που θα επεξεργαστεί τις έννοιες αυτές για να ετοιμάσει ε, της δευτερογενής πράξης στο μέλλον για το ετερογενές υλικό. Τώρα για τους κλόνους. που αναφέρονται στην έκθεση της κυρίας Αγιούζο και υπογραμμίστηκαν ιδιαίτερα. Εδώ θέλουμε να πούμε ότι η καταχώρηση των κλώνων ήδη αποτελεί πρακτική σε ορισμένα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κάποιοι κλόνοι που, είναι, που υπόκεινται ε, σε ε, ε, κάποια ιδιαίτερα κριτήρια επιλογή ή υπάρχουν σε ορισμένες περιφέρειες. Εδώ θα πρέπει να γίνεται καταχώρηση όπου αυτό ε, πρέπει ε, να γίνεται, μπορούμε να το συζητήσουμε και να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Για τους ελέγχους, επιθεωρήσεις, δοκιμές, ε, για την διαπίστευση, για την πιστοποίηση και τις επιχειρήσεις. Εδώ υπάρχει ένα σύστημα δύο επιπέδων. Για να μπορούν οι επιχειρήσεις να κάνουν πιστοποίηση θα πρέπει πρώτα να ε, εγκριθούν από την αρμόδια αρχή και μετά η αρμόδια αρχή θα κάνει έναν έλεγχο η ίδια στον, στους πιστοποιημένους ε, επιχειρηματίες για να διαπιστώσουν ότι εξακολουθούν να συμμορφούνται προς τις απαιτήσεις. Ανεξάρτητα από αυτούς τους ελέγχους θα, γίνουν, θα γίνει ένα ποσοστό ελέγχων με βάση την επικινδυνότητα θα γίνονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα ή ανάλογα με την πιθανότητα μη συμμόρφωσης του υλικού με τις απαιτήσεις του κανονισμού. Εις επίμετρον, αν οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν μόνοι τους αυτή τη δραστηριότητα υπό επίσημη εποπτεία, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να κληθούν οι αρμόδιες αρχές να αναλάβουν αυτά, αυτούς τους ελέγχους και αυτές τις ε, διαδικασίες. Αυτό το θέμα είναι ανοιχτό. Μπορεί να τα αναλάβουν αυτά οι αρμόδιες αρχές. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η συγγήτρια έχει τέλος το λόγο. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα όσα είπατε. Πολλά από αυτά τα συμμερίζομαι. Σε αυτό το θέμα της αποπομπής της πρότασης, πράγματι, αυτή την πρόταση δεν τη ζήτησε κανείς. Κάποιοι ζήτησαν τροποποίηση της, για, τροποποίηση της ισχύωσης νομοθεσίας για να προσαρμοστεί, αλλά κανείς δεν ζήτησε καινούρια πρόταση σε τόσο ετερογενείς και διαφορετικούς μεταξύ τους τομείς. όπως για παράδειγμα το δασικό υλικό ε, που πολλοί το ήθελαν σε διαφορετικό κείμενο. Τώρα, τους ορισμούς πρέπει να τους ε, βελτιώσουμε. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε παράλληλες αγορές διότι το εμπόριο ε, σπόρων και φυτών φυτορίου βρίσκεται στα χέρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τους κλόνους, η πρόταση κάνει, έχει, περιλαμβάνει μια, ένα ορισμό που συμπίπτει με τον ορισμό της, ε, ε της Παγκόσμιας Ένωσης Προστασίας ε, Φυτών και Σπόρων. Όμως μετά, μέσα στην νομοθεσία αναφέρεται η ύπαρξη διαφόρων γενοτύπων, διαφορετικών γενοτύπων στην ίδια ποικιλία και που μπορούν να ε, ε διαχωριστούν επιλεκτικά. Για τους κλόνους έχουμε δύο ετικέτες, έχω εδώ δύο ετικέτες πιστοποιημένων φυτών. Το φυτογενομικό διαβατήριο λέει κοινό όνομα, βοτανικό όνομα, ε, ποικιλία και κλόνος. Υπάρχουν, ε, ε, υπάρχουν ε, ποικιλίε, για παράδειγμα τσαμπέλου, ή, φυτά που ανοίγουν στην ίδια ποικιλία και έχουν διαφορετικούς κλόνους. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να μην συμπεριλάβουμε τους κλόνους εδώ, πολύ δε περισσότερο που εφαρμάζουμε την ομοθεσία σε κάτι που δεν είναι ακριβώς κλόνος. Οπότε το πιο λογικό θα ήταν να αποσυρθούν οι κλόνοι από αυτό το νομοθετικό κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει προθεσμία για την κατάθεση 10 Δεκεμβρίου. 22-23 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Γεωργίας η ψηφοφορία θα γίνει Φεβρουάριο-Μάρτιο και ίσως ε, στα πλαίσια αυτής της θητείας θα πάει να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Τώρα θα ψηφίσουμε το απόγευμα στις 3. Καλό διάλειμμα, καλή όρεξη και συνεχίζομαι ακριβώς στις 3 με τις ψηφοφορίες και την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων.